Good morning. I will... Καλημέρα. Θα αρχίζω να μιλάω πορτογαλικά. Τώρα βάλτε τα ακουστικά σας. Okay, thank you. Good morning. Το πρώτο σημείο της ε, ημερησίας διατάξεως είναι οι ανακοινώσεις της Προεδρού. Έχω μία, ένα κακό νέο να σας κοινοποιήσω, ίσως ε, το ξέρετε ήδη, η κυρία Σφένσον, η πρόεδρός μας, ανακοίνωσε χτες πώς παρετείται από τη θέση της για λόγους υγείας. Βάσει του εσωτερικού κανονισμού, η κυρία Ζαρόκα που είναι η πρώτη αντιπρόεδρος θα καταλάβει τη χειρεύουσα θέση μέχρι την εκλογή του ή της ε, νέας Προέδρου ε, της Επιτροπής μας. Στη χθεσινή συνεδρία των συντονιστών αποφασίστηκε να εκδώσουμε ένα ανακοινωθέν τύπου για να ευχαριστήσουμε εξ ονόματος ολόκληρης της Επιτροπής ε, την κυρία Σβένσον για τις εργασίες της, για την αφοσίωσή της και για όλες ε, τις προσπάθειες ε, που έχει κάνει για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και του θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Έτσι έχει κατάσταση λοιπόν. Νομίζω ότι και εσείς θα λυπάστε όπως και εγώ πάρα πολύ, όχι μόνο διότι η κυρία Σβένσον με εξαιρετικό τρόπο ε, κατήχε την ε, θέση και το ρόλο της Προέδρου, αλλά ε, και για τους λόγους που την οδήγησαν ε, στην παρέτηση. Ε, ταχύτατη ανάρρωση θα της ευχηθώ και ε, ευελπιστούμε ότι σύντομα θα την ξανασυναντήσουμε όπου και να είναι στο Κοινοβούλιο, στη Σουηδία, οπουδήποτε. Τέλος πάντων, τούτου λεχθέντος ελπίζω να περάσατε όμορφα στις διακοπές σας. Καλή επιστροφή ε, σε όλους. Έχουμε εντατικές ε, εργασίες που μας περιμένουν. Ελπίζω να έχετε γεμίσει τις ε, μπαταρίες σας. Ελπίζω όλοι τα μέλη της Επιτροπής, Ιδιερμηνής να πέρασαν ωραία στις διακοπές τους. και να έχουν όλοι νέα ενέργεια και κυρίως βούληση για να εργαστούν σκληρά. Δεύτερο σημείο της ε, ημερησίας διάταξης είναι η έγκριση του σχεδίου ημερησίας διατάξεως. Έχουμε την έκθεση της αντιπροσωπείας ε, που πήγε στο Ζαγκρέπ. Θα το ε, εξετάσουμε ε, μετά στο σημείο 10. Το σημείο 11 που είναι η έκθεση της κυρίας Σβένσον για, την, για το mainstreaming στις εργασίες του Κοινοβουλίου θα αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση. Και Επίσης, στη χθεσινή του συνεδρίαση, οι συντονιστές αποφάσισαν να ζητήσουν από την κυρία Ζαρόγκα να αναλάβει εκείνη την έκθεση της κυρίας Σβένσον, ε, δεδομένου το ότι είναι η πρώτη αντιπροέδρος της Επιτροπής και θα αντικαταστήσει την κυρία ε, Σβένσον, ε, θα ασκήσει την Προεδρία μέχρι την εκλογή του ή της νέας Προέδρου. Νομίζω ότι μπορεί να εγκριθεί το σχέδιο με αυτή την μικρή αλλαγή που προανέφερα. Η κυρία Φιγκυρέιδο έχει ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να ευχηθώ καλή επιστροφή σε όλους μετά ε, από τις διακοπές και να προσυπογράψω όλα αυτά που είπατε. Εχθές στη συνεδρίαση των συντονιστών τονίσαμε ε, πόσο σημαντικό είναι να χειριστούμε σωστά ε, το θέμα αυτό της ασθένειας της Προέδρου μας, ε, της κυρίας Βένσον. Φυσικά συμφωνώ με όλα όσα είπατε αλλά θα ήθελα και ως μέλος της ε, πολιτικής της ομάδας ε, και ε, με την ιδιότητα της φίλης και της συνεργάτηδας εδώ και χρόνια στο Κοινοβούλιο θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τον σημαντικότατο ρόλο που έχει διαδραματίσει η φίλη μας η κυρία Εύα πρίτε Σβένσον στον τομέα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών και της πρόθεσης της ισότητας των δύο φίλων να επενέσω την αφοσίωσή της ε, όχι μόνο ως πρόεδρος της Επιτροπής μας γιατί προήγαγε ε, και καθιστούσε πιο όρατο το έργο της Επιτροπής μας όχι μόνο στο Κοινοβούλιο αλλά και σε άλλες χώρες ε, όπως και στη χώρα μου όπου μετέβει με πανελειμμένα ε, υπερασπιζόμενοι πάντοτε τις ίδιες αρχές, δηλαδή την υπεράσπιση ε, των δικαιωμάτων των γυναικών ως επιτοπλίστων. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστη η κατάσταση και θα ήθελα να σε ευχηθώ ταχύ ανάρρωση και να την ευχαριστήσω ειλικρινέστατα για όλη τη δουλειά που έχει κάνει και να την επενέσω για την προσήλωσή της ε, στο έργο της εδώ στο Κοινοβούλιο και όλος ιδιαίτερα στην Επιτροπή μας. Την ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Φιγκυρέντο. Τώρα θα περάσουμε στο σημείο 3. Άλλες ανακοινώσεις της Προέδρου. Θέλω να σας ενημερώσω ότι αύριο από τις 6 παρατέταρτο μέχρι τις 6.30 ε, ε, θα κάνουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα ακούσουμε την παρουσίαση της κυρίας Βιλία Μπαστό ε, για το, την έκθεση σχετικά με την εμπορία ανθρώπων ε, για παρελθούς και μελλοντικέ εργασίες και μια έκτατη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στο Στρασβούργο στις 15 Σεπτεμβρίου από τις 8.30 μέχρι τις 10.30 για να ε, προβούμε στην ψηφοφορία κάποιων γνωμοδοτήσεων. που πρέπει επιγόντως να ψηφίσουμε. Σημείο 4. Έγκριση των πρακτικών συνεδριάσεων ε, των, ε, της 20 Απριλίου, 14 και 15 Ιουνίου. Έχετε τα στοιχεία στους φακέλους σας. Αν ε, μέχρι το πέρας της συνεδρίασης δεν προβάλλεται ενστάσεις, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων. Σημείο 5. Ανακοινώσει της Προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών. Στις 13 ε, Ιουλίου ελήφθησαν αποφάσεις από τους συντονιστές και τις έχετε στο φάκελό σας. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Σημείο 6 τώρα. Ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας μαζί σας. Ένα λεπτό να βρω και τη δική μου. Ora, o primeiro. O primeiro assunto το πρώτο σημείο είναι η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο. Η συγγήτρια, η κυρία Ματέρα, έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλημερίζω όλες τις συναδέλφους. Ήθελα να διευκρινίσω κάποια σημεία τα οποία καθόρισαν και τον κατάλογο ψηφοφοριών και τον δικό μου αλλά και της πολιτικής μου ομάδα. Ήθελα να κάνω τις διευκρινήσεις αυτές αλλά δεν θα ήθελα να ξαναξεκινήσει η συζήτηση και δεν θα ξαναρχίσει φυσικά η συζήτηση. Δράτω με τις ευκαιρίες και τις παρουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα που δεν ήταν εδώ στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω κάποια σημεία ε, τα οποία ήθελα να διευκρινίσω ως συντάκτρια για τα θέματα προπολογισμού. Όσον αφορά το θέμα Progress, ήθελα να προβλέπουμε τα ίδια κονδέλια που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο ε, κρίσης οικονομικής ε, και κρίσης στον τομέα της απασχόλησης είναι καλό να τηρήσουμε τους στόχους που έχουμε προκαθορίσει στον τομέα της εργασίας, των κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων ευκαιριών. Όσον αφορά όμως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ζήτησα αύξηση κατά 1 εκατομμύριο ευρώ σε πληρωμές ε, για την ε, τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σε σχέση με το ποσό που είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι θεωρούμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα να συσταθεί μια ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου που θα μπορούσε να επικεντρωθεί σε στόχους που αφορούν την ισότητα φύλων μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία και βιώσιμη ανάπτυξη. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα Δάφνη, το οποίο ε, είναι αφιερωμένο στην καταπολέμηση της βίας, θα ήθελα να έχουμε το ίδιο επίπεδο ε, κονδυλίων με το 2010. Θεωρώ ότι αυτό είναι ικανή και αναγκαία θήκη. για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προγράμματα τα οποία ε, αποτελούν αντικείμενο της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά και γιατί θα πρέπει ε, να επικεντρωθούμε και στην άφηξη νέων πόρων, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον ίδιο, ίσως και καλύτερο τρόπο. με λοιπόν της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τους ζητήσω, αν μπορούμε να τους ακούσουμε στη συνέχεια, πώς θεωρούν ότι μπορούν να ε, μειώσουν τις δεσμεύσεις υποχρεώσεων στο πρόγραμμα Δάφνη, χωρίς να υπάρχουν συνέπειες στις εργασίες του ίδιου του προγράμματος και στη βία κατά των γυναικών, των παιδιών και των πιο ευάλωτων ατόμων. Τέλος, για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα ε, των Φύλων στο Βίλνιους, θεωρώ ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ίδια χρηματοδότηση με το 2010. Ήρθα σε άμεση επαφή και με το Ινστιτούτο και υπάρχει ανάγκη για νέους πόρους Ιδίω όσον αφορά τις ε, δαπάνες που αφορούν την ενοικίαση νέων γραφείων, διότι η κυβέρνηση της Λιθουανίας δεν ε, θα τους εκχωρεί πλέον δωρεάν ε, τα γραφεία τα οποία χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το Ινστιτούτο του Βίλνιος. Από το Δεκέμβριο του 2011 πάβει αυτή η δωρεάν χορήγηση. Επομένως χρειάζονται επιπλέον κονδύλια για να ενοικιάσουν νέους χώρους για το Ινστιτούτο, για να στεγαστεί το Ινστιτούτο και επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει και νέο προσωπικό για να μπορέσουν να αφοσιωθούν στα προγράμματα που τους απασχολούν ε, εδώ και αρκετά χρόνια. Ζητώ λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση κάποιες εξηγήσει για τη μείωση του προπολογισμού του συγκεκριμένου Ινστιτούτου, το οποίο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ πόρους αυτή τη στιγμή. Όπως σας είπα και εισαγωγικά, δεν θα ήθελα να ξαναξεκινήσει η συζήτηση αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή είναι παρούσα εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έθεσε αυτές τις και θα ήθελα ε, η Πρόεδρος να μου επιτρέψει να ακούσω την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ζητήματα που έθεσε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ματέρα. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία, ένα λεπτό. Σκέτσκο. Το παρέφθυρα προφανώς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε Ευχαριστώ την εισηγήτρια και τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Γυναικών που έδωσαν την ευκαιρία στην Κομισιό να παρουσιάσει σχόλια για τις δημοσιονομικές τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του 2012. Όπως σημείωσε η εισηγήτρια, προτείνω να διευκρινίσω τα ζητήματα που έθεσε η Επιτροπή σχετικά με το Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων ε, ε, και την ισότητα στο φύλλο στα προγράμματα Progress και Δάφνη. Καταρχήν, εις ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, το σχέδιο προϋπολογισμού της Κομισιόν του 2012 ε, έχει σχέση και στηρίζεται στο δημοσιονομικό προγραμματισμό. Όλες οι υπηρεσίες ε, έλαβαν υπόψη το πλεόνασμα από το προηγούμενο έτος κατά το σχέδιο προϋπολογισμού του 2012. Έτσι λοιπόν η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ινστιτούτο αυτό για το 2012 είναι 7,82 εκατομμύρια ευρώ. 1,84 εκατομμύρια ευρώ από αυτά προέρχεται από το πλεόνασμα του 2010. Έτσι εξηγείται ότι 2,98 ε, εκατομμύρια ευρώ ζητήθηκαν από τον προϋπολογισμό του 2012. Η πρόταση της Κομισιόν λοιπόν ευθυγραμμίζεται με το αίτημα του Ινστιτούτου και επίσης ε, είπαμε να ε, χωριστούν όπως είχε προτείνει το Ινστιτούτο οι γραμμές 1 ε, και 2 του προϋπολογισμού. Έτσι λοιπόν το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2012 έλαβε υπόψη όλα τα κόστη που έχουν να κάνουν με το μίσθωμα. Ε, συνεπώς η Κομισιόν δεν περιέκοψε την επιδότηση του Ινστιτούτου για το 2012, η πρόταση της Κομισιόν σεβάστηκε απόλυτα το δημοσιονομικό προγραμματισμό για το 2012 και αντικατοπτρίζει τα αιτήματα του Ινστιτούτου. Όμως, εις ό,τι αφορά το προσωπικό του Ινστιτούτου για το 2012, το Ινστιτούτο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησαν ε, τρεις ε, νέες προσωρινές θέσεις σύμφωνα με τη νομική βάση και τρεις ε, επισυμβάσει θέσεις. Αυτές οι θέσεις δικαιολογούνται απόλυτα γιατί το Ινστιτούτο είναι σε μια κέρια πρώτη φάση δημιουργίας του ε, όμως ε, ε κόπηκε μία θέση προσωρινή. Αυτό περιορίζει και υπονομεύει τη δυνατότητα που έχει το Ινστιτούτο να ανταποκριθεί στην εντολή του. Κατά δεύτερο λόγο, εις ό,τι αφορά το πρόγραμμα Progress, το σκέλος που αφορά την ισότητα των φύλων για το σχέδιο προϋπολογισμού 2012, το Συμβούλιο περιέκοψε τις πιστώσεις πληρωμών κατά 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Κατά συνέπεια, η σχέση ε, πληρωμών προς υποχρεώσεις από το 80% ε, στην πρόταση της Κομισιόν έπεσε στο 63% στην τροπολογία του Κοινοβουλίου. Αυτό θα μπορούσε να ε, υπονομεύσει το, την υλοποίηση του προγράμματος. Τέλος, εις ό,τι αφορά το ζήτημα για την ε, μείωση των ε, κονδυλίων για το πρόγραμμα Δάφνη, η Κομισιόν πρότεινε στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2012 17,5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο ποσό ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τον αρχικό δημοσιονομικό προγραμματισμό, όμως ε, συγκρίνοντας τα ποσά για το 2011 και το 2012 έχουμε μείωση κατά 2,5 εκατομμύρια. Αυτή η μείωση εξηγείται από το γεγονός ότι στην δημοσιονομική διαδικασία του 2011 η αρχή του προϋπολογισμού μείωσε ε, του 2011 από 17,6 εκατομμύρια ε, αύξησε συγγνώμη, από 17,6 σε 20 εκατομμύρια. Άρα, συνεπώς, δεν υπάρχει περικοπή στα κονδύλια του 2012 όπως προβλέπει ο δημοσιονομικός προγραμματισμός για το πρόγραμμα Δάφνη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Ματέρα, θέλετε το λόγο μετά από αυτή την παρέμβαση, όχι. Ωραία, θα περάσουμε λοιπόν στη ψηφοφορία. Πρώτη τροπολογία. 6201 υπέρ παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 6202 πάλι της κυρίας Ματέρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 6203 της κυρίας Ματέρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 η 20 της κυρίας Ματέρα επίσης υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Τροπολογία 62-21 της κυρίας Παρβάνοβα. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Α. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Α. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6209 της κυρίας Ματέρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 6210 της κυρίας Ματέρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 6222 της κυρίας Φιγκυρέιντο υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62.00. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 62.22. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας. Απορρίφθηκε. 62.00 κυρίας Ματέρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62.23 της κυρίας Φιγκυρέιντο. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Επαλήθευση παρακαλώ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίστε. Πέρας. Απερίφθη. 62-24 πάλι της κυρίας Φιγκυρέιντο, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 62-11 τώρα της κυρίας Ματέρα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 62-25 της κυρίας Φιγκυρέιντο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62-12 της κυρίας Ματέρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62-26 της κυρίας Φιγκυρέιντο υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 62-13 της κυρίας Ματέρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62-30 της κυρίας Ματέρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62-15 Ματέρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62-16 ματέρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62-17 ματέρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62-18 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62-19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και θα ολοκληρώσουμε έτσι την ψηφοφορία αυτής της εκνομοδότησης τον Οκτώβρη θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών 6 με 8 Οκτωβρίου. Συγχαρητήρια στην κυρία Ματέρα. Σημείο 7. Θα περάσουμε τώρα στην ε, ψηφοφορία του σχεδίου γνωμοδότησης για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της ε, φτώχειας και του κοινωνικού ε, αποκλεισμού. Η κυρία Ζαμπόσκα είναι η συγγετριά μας. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω παρατηρήσεις να κάνω. Θέλω να ευχαριστήσω μόνο όλους τους συναδέλφους για τις τροπολογίες. Προσπάθησα άλλωστε να τις λάβω όλες υπόψη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Ζαμπόρουσκα. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογίες 20 ε, και 21 ομού γιατί είναι ταυτόσιμες υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 25 υπέρ, κατά επαλήθευση παρακαλώ, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίθηκε. 26 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 29 υπέρ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 Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 43. Υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 44 και 45 είναι ταυτόσιμες. Ε, μαζί υπέρ. Κατά. Απόχες Νομίζω ότι απορρίπτονται, αλλά θα κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκαν. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 47 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές Ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. 49. Καταπίπτει. 51 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ Ζητάτε επαλήθευση για την 50 παρακαλώ Πέρας Εγκρίθηκε 11 Μήπως θα μπορούσαμε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 Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε ηλεκτρονική επαλήθευση. Παρακαλώ ψηφίστε. Για το δεύτερο τμήμα της 17, έτσι. Πέρασε ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε όντως. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά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 Εγκρίθηκε με 31 ψήφους υπέρ και μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Ζαμπόσκα. Vamos passar ao ponto 8 Σημείο 8 τώρα. Οι τροπολογίες για το τέταρτο φόρουμ υψηλού επίπεδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Η κυρία Κρετού είναι η συγγήτρια. Δεν ξέρω αν θέλει το λόγο. Όχι. Ας ψηφίσουμε τότε. Μπορούμε να τις ε, ψηφίσουμε ομού τις τρεις αυτές τις τροπολογίες ή υπάρχουν αντιρρήσεις. Ωραία, θα ψηφίσουμε λοιπόν και για τις τρεις υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται ομόφωνα συγχαρητήρια στην κυρία Κρέτσου. Και τώρα θα ζητήσω από την Αντιπρόεδρο να με αντικαταστήσει, διότι θα ψηφιστεί η δική μου γνωμοδότηση και θα ήθελα να μιλήσω. Και γι' αυτό θα πρέπει κάποιος να με αντικαταστήσει. Κυρία Σατιέ, παρακαλώ, Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή στο σημείο 9 την έκθεση πρόοδου για το θέμα των αδειών μητρότητας και υπάρχει μια προφορική ερώτηση την οποία προτείνει η κυρία Στρέλα. Το Κοινοβούλιο θέτησε την ε, θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Οκτωβρίου του 2010 όσον αφορά την άδεια μητρότητας, αλλά το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα υιοθετήσει επίσημη θέση για το θέμα αυτό. Στη διάρκεια της τελευταίας του συνεδρίασης, οι συντονιστές ζήτησαν από την εισηγήτρια να προτείνει μία προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο για να δούμε πώς έχει η κατάσταση προόδου του συγκεκριμένου ζητήματος. Η προφορική ερώτηση θα ψηφιστεί στην ε, συνεδρίασή μας σήμερα εν ώψη της ε, Ολομέλειας ε, του Σεπτεμβρίου, της πρώτης Ολομέλειας του Σεπτεμβρίου. Προτείνω λοιπόν να δώσουμε απευθεία το λόγο στην κυρία Στρέλα προκειμένου να μας παρουσιάσει την προφορική ερώτηση και να μπορέσουμε στη συνέχεια να κάνουμε τη συζήτηση. Όπως ε, είπε ήδη ε, προεδρεύουσα, έχουμε αντιμετωπίσει κάποιες αντιξοότητες ε, σε αυτό το τομέα και η τελευταία σχετίζεται με την έλλειψη θέσης από πλευράς του Συμβουλίου σχετικά με την ε, εγκεκριμένη από το Κοινοβούλιο θέση ήδη πέρσι ε, τον Οκτώβρη. Ω εκ τούτου αποφασίστηκε στη συνεδρία των συντονιστών πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές ότι θα υποβάλαμε μία προφορική ερώτηση με αίτημα για προφορική απάντηση, δηλαδή με συζήτηση στην Ολομέλεια. Αποστήλαμε μέσω των συντονιστών αυτό το αίτημα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι διάφορες πολιτικές ομάδες αντέδρασαν και κατέθεσαν τροπολογίες. Εγώ δέχθηκα όλες τις τροπολογίες που υπευλήθησαν. Δέχομαι την τροπολογία της ΓΚΟΕ για την ε, παράγραφο 5 διότι υπάρχει μία συνοχή. Δηλαδή, ε, αναφερόμαστε σε μία προθεσμία, μία καταληκτική προθεσμία ε, σχετικά με όλε όλες τις προτάσεις που έχω συμπεριλάβει στην έκθεσή μου η οποία έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο μέχρι το 2020. Ε, δηλαδή μέχρι ότου η στρατηγική ε, Ευρώπη 2020 ε, εφαρμοστεί και άρα όλοι οι στόχοι που σχετίζονται με αυτή την πολιτική, με αυτή τη στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να δημιουργήσουν προϋποθέσεις τέτοιες ώστε όλα τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τα εν λόγω μέτρα του τέστη ε, θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη διαλλακτικότητα ε, δεδομένης της κατάστασης που βιώνουμε, η οικονομική, χρηματοπιστωτική, κοινωνική κρίση. Όλοι γνωρίζουμε φυσικά πολύ καλά την κατάσταση που επικρατεί και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η κρίση στα επιμέρους κράτη-μέλη. Γι' αυτό ε, και προτείνω να υιοθετηθεί η μεταβατική ρήτρα, η περίφημη ρήτρα Πασερέλ και με τα μέτρα που θα υιοθετήσουμε θα εφαρμοστεί σταδιακά αυτό, αλλά θα περατωθεί η διαδικασία το 2020. Θεωρώ ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από το να πούμε ότι κατεπηγόντως πρέπει να υιοθετηθούν όλες οι ρήτες. Ε, είναι, είναι πιο διαλεκτικό να πούμε ότι μέχρι το 2020 θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί αυτά τα μέτρα. Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία. Ε, ήρθα σε επαφή με την Πολωνική Προεδρία και αυτή τη βδομάδα έχω άλλη μια επαφή, άλλη μια σύσκεψη μαζί τους. Επίσης ήρθα σε επαφή με την Επίτροπο Ρέντινγκ ε, σε άτυπο επίπεδο. Είχαμε διάφορες άτυπες επαφές ε, με στόχο την εξέβρεση λύσεων για να πεμπλακεί ε, η όλη διαδικασία και για να βρούμε μία λύση που αντιστοιχεί και στην πραγματικότητα αλλά και στις ε, προσδοκίες ε, των γυναικών, των, οικογενειών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό ζητώ από την Επιτροπή μας να εγκρίνει αυτή την προφορική ερώτηση με έτοιμα προφορικής απάντησης για να διαπιστώσουμε ποια είναι η επίσημη θέση του Συμβουλίου και όπως σας είπα η Πολωνική Προεδρία δείχνει ιδιαίτερη δέσμευση και αφοσίωση για αυτό το θέμα. Παρόλα αυτά χρειαζόμαστε ε, τη θέση του Συμβουλίου και η θέση του Συμβουλίου διαφέρει κατά τι από την εκπεφρασμένη βούληση της Πολυνικής Προεδρίας. Ε, το Κοινοβούλιο όμως εμείς θέλουμε να, ε, έχει, να γνωρίζει την επίσημη θέση του Συμβουλίου. Ποιες είναι οι επίσημες προθέσεις λοιπόν του Συμβουλίου σε αυτό το θέμα σε σχέση με τις προτάσεις που υιοθετήθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν. Ευχαριστούμε την ηθικήτρια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα την ανταλλαγή απόψεων. Η κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην πολιτική θα πρέπει να γνωρίζουμε αυτό που λένε οι μεγάλοι οι Γάλλοι φιλόσοφοι ότι ό,τι είναι υπερβολικό είναι ανούσιο. Εμείς υιοθετήσαμε μία υπερβολική θέση όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της άδειας μητρότητας και το Συμβούλιο προφανώς αποφάσισε ότι δεν έχει καμία σημασία και δεν θα το συζητήσει, δεν θα συζητήσει επί τη βάση μιας υπερβολικής θέσεως. Δώσαμε μια μάχη για μια πιο ρεαλιστική θέση, πιο λογική, η οποία θα μπορούσε ίσως να ε, τύχει και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου, αλλά το Κοινοβούλιο είπε ότι ήθελε 20-22 παραπάνω και τώρα η αντίδραση του Συμβουλίου είναι αυτή που γνωρίζουμε. Διότι ήδη και στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας μας είχαν πει, γιατί εγώ είχα πολλές επαφές με την Ισπανική Προεδρία για το δικό μου το ζήτημα το οποίο πέρασε. Η Ισπανική Προεδρία λοιπόν μας είχε ήδη πει ότι αν το κάνετε αυτό, αν ψηφίσετε αυτή την έκθεση με αυτές τις υπερβολές, το Συμβούλιο δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα και ούτε και οι άλλοι θα κάνουν τίποτα, διότι η θέση μας είναι υπερβολική. Τώρα προσπαθείτε από την πίσω πόρτα, πόρτα μέσω μιας προφορικής ερώτησης να ξανανοίξετε αυτό το ζήτημα με το Συμβούλιο είναι τραγελαφικός αυτός ο τρόπος που προσπαθούμε να προχωρήσουμε τις εργασίες μας. Ποτέ δεν έγινε αυτό έτσι. Υπάρχουν διαδικασίες που μπορούμε να καθορίσουμε. Γιατί να συζητήσει το Συμβούλιο μαζί σας. Έχετε μία θέση και έχετε αιμονή με αυτή την υπερβολική θέση. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι αστείος αυτός ο τρόπος. Προσπαθούμε από την πίσω πόρτα τώρα να επανορθώσουμε τη ζημία που προκαλέσατε υιοθετώντα αυτή την υπερβολική σας θέση και εγώ προσωπικώς δεν συμφωνώ. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ. Η κυρία Φιγκερέιδο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε προηγούμενες συνεδριάσεις, πριν από τις καλοκαιρινές μας διακόπες, αποφασίσαμε να υποβάλουμε αυτή την προφορική ερώτηση. Ε, η Αντίτα Στρέλα παρουσίασε τα δεχτούν αυτά που προτείνουμε τα κράτη-μέλη και στο κάτω-κάτω τη γραφής το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο αποτελείται από τρία τμήματα από ό,τι γνωρίζω. Εκείνο της Κομισιόν, του... τα ε, ε, θεσμικά όργανα είναι τρία και θα πρέπει να συνεργάζονται. Ε, μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες στη θέση του Κοινοβούλου και εμείς θα αντιταχθούμε γιατί όπως είπαν οι συνάδελφοι εκπροσωπούμε τα κράτη-μέλη και εμείς. Ίσως λοιπόν το θέμα πρέπει να το αφήσουμε, να το ξαναδούμε, να το αποδυναμώσουμε λίγο για να γίνει δεκτό. Είναι θέμα απασχόλησης. Εμείς πρέπει να επικεντρωνόμεθα σε πράγματα που μπορούμε να επηρεάσουμε και να μην ε, επιμένουμε σε πράγματα που δεν έχουν προοπτική επιτυχίας. Νομίζω ότι θα με υποστηρίξουν και οι διαφωνούσες συνάδελφοι εδώ. Σας ευχαριστούμε η κυρία Μπάουερ. Μα εμείς ε, θα προβάλλουμε βέτο έτσι μέχρι τελευταία στιγμής. Ευχαριστώ. Μια σύντομη παρατήρηση. Δεν υπάρχει πρόθεση να επαναλάβουμε τις συζητήσεις και αυτά που κάναμε πριν από ένα χρόνο. Είμαι βεβαία ότι αν συνεχίσουμε να λέμε ότι το λιγότερο θα είναι περισσότερο, ε, το, αν το λέγαμε, τότε η οδηγία θα ήταν σε ισχύ. Εν πάση περιπτώσει, έχω την εντύπωση ότι επειδή ενημερώθηκαν, ενημερώθηκε και το Συμβούλιο για το θέμα, αυτό δεν είναι τόσο κακό. Θυμίζω ότι η διατήρηση της οδηγίας πάνω στο, στη βάση του, της υγείας και της ασφάλειας θα ήταν πιο λογικό. Μπορεί κάποιος να ηρωοποιηθεί με από ε, κάποιο λαϊκισμό ανεδαφικό, ενώ είναι δύσκολο να βρεθεί μια πραγματική ισορροπία σε τέτοιου είδους περιπτώσεις και θέματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να ε, τεθεί το θέμα στο Συμβούλιο, αφού δεν σημειώθηκε μέσα σε ένα χρόνο καμία πρόοδος και δεν δόθηκε μια ε, ενημέρωση σε σχέση με την πορεία του θέματος αυτού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς ε, για τα τυπικά. Η προφορική ερώτηση θεωρώ ότι είναι εξαίρετη μέθοδος για να παραμείνει ένα θέμα ανοιχτό και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση από αυτού. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι προφορικές ερωτήσεις και νομίζω ότι καλώς ε, χρησιμοποιούμε προφορική ερώτηση σε αυτή την περίπτωση. Δεύτερον, ω Ευρωβουλευτή αλλά και ω εμπειρογνώμονα σε διεθνέ ε, δημόσιο δίκαιο να σας υπενθυμίσω το εξή. Πριν από 20 εβδομάδες, από 20 χρόνια συγγνώμη, απαγορευόταν να τεθούν ερωτήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προς μια κυβέρνηση. Θεωρείταν ακατάλληλο και δεν γινόταν. Μετά από πολλή δουλειά και στο θέμα των Ηνωμένων Εθνών πριν από 20 χρόνια ο μόνος τρόπος να θέσει κάποιος ε, μία ερώτηση ήταν ε, να υπάρχει κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γινόταν μία μυστική διαδικασία. Πλέον έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Υπάρχουν ε, καθημερινώς θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρούμε ότι είναι κάθε δικαίωμα του Κοινοβουλίου να θέτει ερωτήσεις προς τις κυβερνήσεις και τους φορείς των Ηνωμένων Εθνών. Και πώς επετέφθη αυτή η αλλαγή μέσω του έργου των βουλευτών παγκοσμίων Ταμείο σε όλες τις χώρες. Και νομίζω ότι το να λέμε ότι εάν όλες οι κυβερνήσεις λένε όχι στο Συμβούλιο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ένα θέμα, δεν είναι απάντηση. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη αποστολή. Ασχολούμαστε με την ισότητα των φίλων εδώ στην Επιτροπή μας και αν υποχωρήσουμε εμείς, ποιος θα υπερασπιστεί αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Εκ. Ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα να λάβω το λόγο, αλλά μετά από τα όσα διεμήφθησαν θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ακουστεί και η δική μας η άποψη. Δύο ερωτήσεις. Μία ως προς τα βασικά. Η ισότητα και η ελεύθερες επιλογές για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευρωπαϊκό ζήτημα κατά την άποψή μας. Δεν είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το άλλο θέμα που ήθελα να θίξω και που αναφέρθηκε είναι ότι εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες. Έχουμε δική μας εντολή, έχουμε δική μας ευθύνη ανεξάρτητα από το τι αποφασίζουν οι κυβερνήσει των κρατών μελών, τι ψηφίζουν και τι παρακολύουν σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν λοιπόν εκπροσωπούμε τη βούληση των πολιτών και τις ανησυχίες των πολιτών και τις ε, τους πολίτες εν γέννη, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα τους πολίτες μας. και στις επικράτειές μας και σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, να θέσουμε το θέμα επιτάπητος προς συζήτηση. Και αυτό ζητούμε μόνον μέσω αυτής της προφορικής ερώτησης. Η τελική απόφαση βέβαια δεν εξαρτάται μόνον από τη θέση μας, αλλά το γεγονός ότι θα πρέπει να συζητηθεί είναι αδιαμφισβήτητο. Και γι' αυτό και υποστηρίζουμε πλήρως την πρόταση της κυρίας Εστρέλα ίσως με κάποιες ε, μικρές τροποποίησεις και κάποιες προσθήκες, αλλά η αρχή είναι ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση, θα πρέπει να συνεχίσει να ενημερώνονται οι πολίτες και να πρέπει να υπάρξει μία λύση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν θα πρέπει να υποτιμούμε το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστούμε κύριε Ρωμέβα. Η κυρία Τόμσεν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε κάτι την αντίληψη που έχουμε περί άδειας μητρότητας. Εγώ προσωπικά ε, ήμουνα σε ένα δανέζικο συνδικάτο στο παρελθόν και λέγαμε ότι η οι κοινωνικοί εταίροι θεωρούν ότι είναι ζήτημα απασχόλησης η άδεια και θα το ξαναπώ σήμερα, είναι θέμα απασχόλησης. Υπόθηκε επίσης ότι είναι θέμα υγείας και ασφάλειας. Η άδεια κατά τη γνώμη είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αυτή την πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η γυναίκα δικαιούται να κάνει ένα παιδί και να πληρώνεται κανονικά και να μην τιμωρείται ε, επιπροσθέτως δηλαδή πέρα από την εγκυμοσύνη και όλες τις δυσκολίες που συνεπάγεται αυτή. Αν ήταν ε, θέμα απασχόλησης, εντάξει, να συμφωνήσω, αλλά οι κοινωνικοί εταίροι δεν συζητάνε για την αποζημίωση και ποιος δικαιούται ή δεν δικαιούται ε, την άδεια μητρότητας. Δεν συζητούν αυτό. Οι εταίροι της αγοράς εργασίας ε, θέλουν η άδεια ε, μητρότητας ε, να λειτουργήσει διαφορετικά και να είναι όμοιροι οι γυναίκε στη διαδικασία. Δεν συμφωνώ. Ε, το Συνδικάτο των Οδηγών Φορτηγών, παραδείγματο χάρη, δεν πιστεύω ότι πρέπει να επηρεάζει την κατάσταση των γυναικών που θέλουν να γεννήσουν ένα παιδί και δυστυχώ σε πολλά κράτη-μέλη η άδεια μητρότητα δεν είναι θέμα απασχόληση, είναι ένα δικαίωμα. Λαμβάνει πλήρη αμοιβή η γυναίκα σε χώρε όπω στην Πορτογαλία Γαλλία παραδείγματο χάρη σε άλλε χώρε. Δεν πρέπει λοιπόν να βλέπουμε του πιο συντηρητικού και αντιδραστικού τι κάνουν. που δεν εξασφαλίζουν δηλαδή την ισότητα των δικαιωμάτων των δύο φύλων, θα πρέπει να προβάλλουμε τις ε, χώρες ε, που έχουν σημειώσει πρόοδο. Και παρακαλώ να παραμείνει έτσι αυτό το θέμα, να είναι ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε κυρία Τόμψεν, ο κύριος Σιμόσκι. Ε, έχει το λόγο. Ε, myślę, że tu nie musimy przekonywać co do poglądów, e, Δεν νομίζω ότι πρέπει να πείσουμε εδώ ένας τον άλλον. Άλλωστε η Επιτροπή μας είναι πολύ ευαισθητοποιημένη σε όλα αυτά τα θέματα παρά τις διαφορές μας. Το ζήτημα είναι αν θα είναι αποτελεσματική η δράση μας αυτή, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της εφορίας που επικρατεί στο Κοινοβούλιο και της πραγματικής κατάστασης. Ποια λοιπόν, ποιος είναι ο σκοπός της πρωτοβουλίας. Εγώ συμμερίζομαι τις προθέσεις. Το ζητούμενο είναι, αν θα συνεχίσουμε τη συζήτηση όμως, καταδεικνύοντας κάτι, αν η Ευρώπη πρέπει να δει πώς παλεύουμε για το ζήτημα αυτό, ποια είναι η γνώμη μας γι' αυτό και ή αν θέλουμε να αποκομίσουμε, να κερδίσουμε κάτι. Το θέμα είναι αν υπάρχει θεσμικό πρόβλημα και το ερώτημα αφορά την αποτελεσματικότητα των δράσεων. Είναι σοβαρό το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να πούμε ειλικρινά ότι όλο αυτό το θέμα αποτελείται από πολλές ε, δυνατότητες και δράσεις για να υπάρξει συμβιβασμός. Αν ασκηθεί βέτο, μπλοκάρονται τα πάντα. Και τώρα διακυβεύεται το κύρος μας, γιατί έχουμε εμείς μια δημοκρατική εντολή και πίσω μας ε, βρίσκονται εκατομμύρια πολίτες. Ενώ στο τέλος δεν θα γίνει τίποτε. Να αντιδράσουμε λοιπόν, αλλά πώς. Όχι έτσι τα πρότυπα για την προστασία των γυναικών και την προστασία της άδεια μητρότητα στην Ευρώπη θα βελτιωθούν ως αποτέλεσμα των δράσεών μας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διάσταση στο, ε, ερώτημα, στο ζήτημα αυτό. Και εμείς θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, Κομισιόν, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο. Γιατί κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχει η δημοκρατική μας εντολή, εμείς κάνουμε τόσες σοβαρές εργασίες και οι κυβερνήσεις που έχουν την, ε, όλη την ισχύ μπορούν να μπλοκάρουν τα πάντα. Το θέμα λοιπόν αυτό της ε, ε, υπερβολής έχει κάποια βάση, γιατί πρέπει να θέσουμε στόχους φιλόδοξους μεν, αλλά στόχους που θα φέρονται και θα βρίσκουν σύμφωνα σε όλες τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι το συζητούμενο. Κύριε Λούλιν. Ευχαριστώ διαδικαστικό, Πρόεδρε ούτε θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι εδώ, ούτε θέμα γοήτρου, ούτε τίποτα. Είναι θεσμικό το ζήτημα. Είμαστε ε, σε περίοδο συναπόφασης, στη διαδικασία συναπόφασης με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Και κατά τη διάρκεια συναπόφασης. Ε, δεν έχουμε τέτοιο προηγούμενο, προφορική ερώτηση με συζήτηση στην Ολομέλεια, ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Ε, εγώ συστήνω να υποβάλουμε μια σχετική ερώτηση στη νομική υπηρεσία για να δούμε αν θα γίνει παραδεκτή ε, η ερώτηση, διότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι επιρροής του Συμβουλίου όλοι ε, είμαστε υπέρ της αναβάθμισης, της βελτίωσης ε, της ε, υφιστάμενης οδηγίας. Αν είχατε δεχθεί τις ε, λογικές ε, προτάσεις που είχαμε κάνει θα την είχαμε ήδη την οδηγία ε, και με μια βελτίωση ίσως όχι 5 ως 6 εβδομάδες αλλά τουλάχιστον 2 ως 4 εβδομάδες. Αν δεν θέλετε λοιπόν να ακούτε τις λογικές προτάσεις να υπομειστείτε τις ευθύνες σας, εσείς ευθύνεστε γιατί εσείς υπερβάλλατε και εξαιτία σας δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτό το θέμα και γι' αυτό το λόγο ζητάω η Επιτροπή μας να ζητήσει γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας ε, αν δηλαδή ε, τη της διαδικασίας συναπόφασης είναι δυνατόν να υποβληθεί η προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια για ε, συζήτηση. Αν θα γίνει παραδεκτό το αίτημα ή αν θα βρεθούμε πάλι σε μια κατάσταση όπου θα απολέσουμε κάθε εξοπιστία. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ε, οι δύο τελευταίοι ομιλητές, η κυρία Ζαμπόσκα πρώτον. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε όντως σε δύσκολη θέση. Η οδηγία αυτή αφορά την προστασία της υγείας των εγγύων γυναικών και των γυναικών μετά τη γέννα Άρα εμείς πρέπει να αναλάβουμε συγκεκριμένη ευθύνη εδώ. Η κατάσταση σήμερα των εγγύων γυναικών σε κάποια κράτη-μέλη δεν είναι η καλύτερη. Η νομοθεσία δηλαδή δεν λαμβάνει υπόψη τη συμβολή των γυναικών στην κοινωνία με τη μορφή συγκεκριμένης οικονομικής αν θέλετε ε, αποκατάστασης ή μέσα από την προστασία της άδεια μητρότητας. Πιστεύω ότι το να θέσουμε μια εκτενή ερώτηση μαζί με τις τροπολογίες που θα υποβάλλουμε στο Συμβούλιο, νομίζω ότι αυτό δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απόλυτα καθαρή. Ε, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια και θα τεθεί μια ερώτηση προς το Συμβούλιο με την έννοια ποια είναι η γνώμη σας, ποια είναι η θέση του Συμβουλίου δηλαδή, πότε θα εγκριθεί η νομοθεσία και δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό να υποβάλλουμε άλλες προτάσεις γιατί ήδη ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα εκεί σε συνάρτηση με τη γνωμοδότησή μας. Και πραγματικά δεν ε, ξέρω τι θα μπορούσε σε αυτό το ζήτημα να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά η λύση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, αποσύρει την πρόταση για να επεξεργαστεί ένα νέο κείμενο, ίσως ε, δεν θα ε, ήταν τόσο κακή ιδέα. Θα μπορούσε αυτό να το δεχτεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Δεν ξέρω λοιπόν μήπως θα έπρεπε το ζήτημα αυτό να το απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και να την ρωτήσουμε τι συνέχεια βλέπει να δίδεται σε αυτή την νομοθεσία. Ε, ρώτηση προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο, χωρίς άλλες ε, τροπολογίες. Αυτό πιστεύω ότι είναι το καλύτερο και αντικατοπτρίζει και την ψηφοφορία που είχαμε στην Ολομέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ζαμπόρκα. Η κυρία Τσέσκοβα είναι η τελευταία ομιλήτρια. Uh, Ευχαριστώ. Πολύ σύντομη θα είμαι. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την άδεια μητρότητας που είναι βασικό δικαίωμα. Μόνο σε προαιρετική βάση μπορεί να τεθεί και όχι υποχρεωτική για αυτό το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, για να ανακεφαλαιώσει, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε μια απάντηση στην παρατήρηση της κυρίας Λούλινγκ. Εξετάσαμε τα έγγραφα και το άρθρο 115 λέει ότι αποφασίζει η διάσκεψη των προέδρων κατά πόσον θα είναι παραδεκτό ή μη παραδεκτό ένα αίτημα. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε εμείς να ψηφίσουμε για την προφορική ερώτηση και κατόπιν η διάσκεψη των Προέδρων θα μπορέσει να αποδεκτεί ή να μην αποδεκτεί ε, την προφορική ερώτηση ε, στην ημερήσια διάταξη. Αυτό προτείνω. Η κυρία Στρέλα τώρα έχει το λόγο, η οποία είναι και η συντάκτρια της προφορικής ερώτησης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα τα σχόλια, διαπίστωσα ότι οι πλήστοι συνάδελφοι υποστηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία, να υποβάλουμε δηλαδή μία προφορική ερώτηση για το Συμβούλιο με συζήτηση. Η συζήτηση που έγινε ε, δεδομένου του αριθμού και της ποιότητας των παρεμβάσεων καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να κάνω και κάποια σύντομα σχόλια. Δεν θα ε, επαναλάβω τώρα όλη αυτή τη συζήτηση και την επιχειρηματολογία γιατί μέσα έχει απασχολήσει σε πολλές συνδυάσεις το θέμα. Θα ήθελα απλώς να σας θυμίσω ότι με τη δημογραφική πρόκληση της Ευρώπης με τα χαμηλά ποσοστά γεννηδικότητας και με όλους ε, με όλα αυτά τα κίνητρα που θα πρέπει ε, να ε, προσφέρουμε για να αυξηθεί η γεννητικότητα καλό θα κάναμε να στηρίξουμε όλα αυτά τα μέτρα. Ε, πρόκειται προφανέστατα για βασικά δικαιώματα η άδεια μητρότητας και η άδεια πατρότητας. Πλην όμως δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι ε, συνιστά βάρος για την κοινωνία η άδεια μητρότητας. Αυτή την οτροπία θα πρέπει να αλλάξουμε ε, και όλος ιδιαιτέρως στους κόλπους του Συμβουλίου. Όπως είπε η κυρία Ζαμπόσκα, η άδεια μητρότητας είναι μια υπηρεσία προς την κοινωνία. λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες ε, που βιώνουμε όλοι, Θεωρώ ότι με αυτήν την ερώτηση αυτό που κάνουμε είναι να επαναλαμβάνουμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Ε, διότι δεν μπορεί η προσωπική μας θέση να υπερακοντίζει την ε, κοινή θέση του Κοινοβουλίου. Οφείλουμε να σεβαστούμε την έκβαση της συνειδητής ψηφοφορίας που έγινε στο Κοινοβούλιο ε, σε όλες τις πολιτικές ομάδες αποτέλεσε ε, το θέμα αυτό αντικείμενο ε, εκτεταμένων συζητήσεων. Είναι αφιλεγόμενο το θέμα και εν πάση περιπτώσει με πλήρη συνείδηση τοποθετήθηκαν όλοι οι βουλευτές στο Κοινοβούλιο και άρα θα πρέπει να δούμε ποια είναι η θέση της Επιτροπής και του Συμβουλίου αντίστοιχα. Αναφερθήκαμε στη ρήτρα Πασερέλ, στη μεταβατική ρήτρα. και προσπαθούμε εδώ να είμαστε πιο διαλλακτικοί, να υποβάλουμε μια πιο ρεαλιστική πρόταση ε, και προτείνουμε να οριστεί αυτή η προθεσμία μέχρι το 2020 θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί όλες οι προτάσεις που έχει ήδη εγκρίνει το Κοινοβούλιο στην θέση του. Ε, τώρα δεν θα αρχίσουμε θεωρητικέ συζητήσει για τη δημοκρατία και ποιοι είναι οι αιρετοί αληθινοί εκπρόσωποι του λαού και ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θα ήθελα να ε, θυμίσω στην κυρία Σινκλέρ ότι εσχάτως και μετά από όλη αυτή την συζήτηση στην ίδια την κοινωνία του Ηνωμένου Βασιλείου ε, προέκυψε μία ε, τροποποιητική πρόταση σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία πηγάζει από ε, τους κανονισμούς του Κοινοβουλίου. Η Πολωνία ε, έχει ήδη τροποποιήσει την νομοθεσία της, ε, το Βέλγιο ακολουθεί μια αντίστοιχη διαδικασία, δηλαδή δημιουργείται ένα κίνημα που αποδεικνύει ότι άξιζε τον κόπο. Όλη αυτή η συζήτηση δηλαδή ε, που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχε επέφερε καρπούς ε, και βοηθά στην ε, αλλαγή της νοοτροπίας καθώς και στην τροποποίηση ε, της κάστοτε εθνικής νομοθεσίας. Η πολιτική είναι η βασίλισσα των συμβαστικών λύσεων. Έτσι λένε αυτοί που μας επικρίνουν. Μάλιστα. Και εμεί ε, θέλουμε ε, να καταλήξουμε σε μια συνενετική λύση με το Συμβούλιο. Πώ λοιπόν θα καταφέρουμε ε, να βαστική λύση μόνο ξανανοίγοντας τη συζήτηση. πώ αγνοώντας τη θέση του Συμβουλίου θα σημειώσουμε η πρόοδο. Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο θα πρέπει να σεβαστεί τη θέση ε, του Κοινοβουλίου, να τοποθετηθεί σε σχέση με τη δική μας θέση, ούτως ώστε από κοινού να απορρευτούμε και να καταλήξουμε σε μια ε, ικανοποιητική για όλους λύση. Ως εισηγήτρια τονίζω ότι ε, προτίθεμαι να συνεργαστώ στενά με τους συντονιστές, με τους σχέδιους με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρόπο ώστε να ε, σημειώσουμε την επιθυμητή πρόοδο και ε, η οδηγία να αναθεωρηθεί το ταχύτερο δυνατόν δύναμη των επιθυμιών, των προσδοκιών των συμπολιτών μας. Φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, την άποψη των κοινωνικών εταίρων και ε, θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις. Δηλαδή, ε, δεδομένων των εξελίξεων πρέπει να αναθεωρηθεί αυτή η οδηγία. Θέλω να συνεργαστώ μαζί σας, θα έχω ανοιχτό πνεύμα, θέλω να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση από κοινού. σας ευχαριστούμε κυρία Εστρέλα. Εκτάκτος ε, θα δώσω το λόγο στην ε, Μαρίνα Γενακουντάκης και μετά όμως ε, θα περάσουμε στην ψηφοφορία, έτσι. Διευκρινιστικά, η Βρετανική κυβέρνηση έκανε εργασίες για την άδεια μητρότητας και δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό που προτείνεται και αυτό που γίνεται είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό πιστεύω τελικά. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε την παράγραφο 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Ένα σχόλιο εκτός μικροφώνου από την κυρία Γιανακουδάκη. Πέρασες ψηφοφορία τώρα. 16 υπέρ, 17 κατά. Απορρίπτεται. Παράγραφος 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση και πάλι άρχεται η ψηφοφορία πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται παράγραφος 5 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία Le vote est clos. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Παραγραφός 7α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 27 ψήφοι υπέρ, 5 κατά και μία αποχή. Σας ευχαριστώ πολύ και ξαναπαραδίδω τα ενία στην κυρία στρέλα Oh, no. Ευχαριστώ πολύ την ε, Αντιπρόεδρό μας, την κυρία Σατιέ, που προείδρευσε ε, το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης. Θα περάσουμε τώρα στο ε, σημείο 14 σχετικά με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Δικαιωμάτων Γυναικών στο Ζάγκρεμπ. Η κυρία Σβένσον απουσιάζει, ε, εκείνη προείδρευσε στην αντιπροσωπεία. Η κυρία Ζαμπρόσκα που ήταν επίσης μέλος της αντιπροσωπείας θα πάρει τώρα το λόγο για να μας ε, ενημερώσει για αυτό το σημαντικό ταξίδι στο Ζάγκρεπ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπατε, στις 16 ε, και 17 Ιουνίου η αντιπροσωπεία της Επιτροπής επισκέφτηκε το Ζάγκρεμπ λίγες μόνο μέρες μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επιορισμένων κεφαλαίων στα πλαίσια της μετά την ολοκλήρωση δηλαδή των διαπραγματεύσεων για ορισμένα κεφάλαια που αφορούν την προσχώρηση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Κροατίας. Ε, τέσσερα ήταν τα μέλη που συμμετείχαν εκτός από την επικεφαλής ε, της γραμματείας μας ε, και την Ίνα Σοκόλσκα από την γραμματεία επίσης όπως και η πολιτική σύμβουλη των σοσιαλιστών και δημοκρατών και της ομάδας των φιλελευθέρων. Νομίζω ότι οι συναντήσεις μας ε, ε, έλαβαν χώρα σε πολύ ψηλό επίπεδο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και σε κυβερνητικό επίπεδο είχαμε συναντήσεις ε, όπως και με εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σε κάθε συνάντηση μιλήσαμε, συζητούσαμε τις διαπραγματεύσεις και την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στην αρχή συναντήσαμε τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Μπελίτη στην Κροατία, ο οποίος μας έδωσε πληροφορίες για όλη την ενταξιακή ε, διαδικασία από την αρχή της και στην πρώτη πρώτου του 2013 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Η παρακολούθηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με αυτά που είχαμε προβλέψει. Η Κροατία συνεχώς επιτηρείται, παρακολουθείται και οι Κροάτες οι ίδιοι θέλουν το monitoring. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι το 2013. Οι μεταρρυθμίσεις κυρίως και η καταπολέμηση της διαφθοράς μας ε, απασχολούν και μας ενδιαφέρουν. Παράλληλα, η ατζέντα σε σχέση με τη δικιά μας επιτροπή αφορά την κατάσταση των γυναικών, την απασχόλησή τους και αυτό αποτελεί επίσης ε, τμήμα του monitoring, του ε, ελέγχου που γίνεται. Η συνάντηση με τους ε, εκπροσώπους της ισότητας των φίλων του Κροατικού Κοινοβουλίου με επικεφαλή στην κυρία Σόμπολ ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και μπορούμε να πούμε ότι η Επιτροπή αυτή ε, συστάθηκε το 2001, έχει 11 μέλη, τόσο γυναίκες όσο και άνδρες και η Επιτροπή αυτή έχει αναλάβει ε, πολλά καθήκοντα, μεταξύ άλλων παρακολουθεί την ε, διαδικασία εφαρμογής της νομοθεσίας Επίσης ε, παρακολουθεί την έγκριση όλων των νομοθετημάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων. Είτε πρόκειται για ποινική η νομοθεσία, η νομοθεσία για το οικογενειακό δίκαιο κατά της βίας μέσα στην οικογένεια, ε, το, στρατηγικό, το πέμπτο στρατηγικό σχέδιο για τις γυναίκες και συμμετέχει επίσης η Επιτροπή στην προετοιμασία των νομοθετημάτων για την παιδεία, την κοινωνική πολιτική, ε, κοινωνικά θέματα, ε, επιχειρηματικέ δραστηριότητες για τις γυναίκες, σχέσεις μεταξύ των ε, δύο φύλων κλπ. Η κυρία Σάμπολ, πρόεδρος της Επιτροπής, μας είπε ότι έχουν ένα πρόβλημα οικονομικό και ότι δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια ώστε να εφαρμόζονται σωστά ε, τα νομοθετήματα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα ε, για τους νόμους υποστήριξη της ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων. Τα προβλήματα νομίζω ότι είναι παρόμοια ε, ως προς αυτό σε όλα τα κράτη. Όλες οι αντιπροσωπείες θεωρούν ότι το οικονομικό πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο πρόσκομα για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Επίσης, ε, Μιλήσαμε, ε, συναντήσαμε και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στη νομοθεσία για τις ποσοστώσεις, γιατί η κροατική νομοθεσία θα πρέπει να προσαρμοστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε το 40% των μελών του Κοινοβουλίου βάσει νόμου να είναι γυναίκες. Ο πρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου θεωρεί ότι μετά την έγκριση του νόμου αυτού η κατάσταση θα βελτιωθεί. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση πραγματοποιήθηκε και με την εκπρόσωπο των πολιτών για την ισότητα. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες παρατηρήσεις που έκανε. Είπε συγκεκριμένα ότι η νομοθεσία θα πρέπει να τροποποιηθεί και θα πρέπει να υπάρχουν τρεις ε, εκπρόσωποι των πολιτών για την ισότητα, για τα δικαιώματα των παιδιών και για τους αναπήρους. Θα πρέπει να συσταθεί ε, ένα ε, μια υπηρεσία ε, στην οποία θα εργάζονται οι τρεις αυτοί. Από την άλλη πλευρά είναι κατανοητό ότι η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο πρέπει να χρησιμοποιεί και θέλει άλλωστε να χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα τα κονδύλια μέσα από την μείωση της γραφειοκρατίας. Από την άλλη, συνήγοροι των πολιτών ε, συμφωνούν και μας διαβεβαίωσαν ότι θα διατηρηθούν τα απαραίτητα χαρτοφυλάκια και οι υπεύθυνοι θα εξακολουθήσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Απλώς θα ενταχθούν σε μία ε, υπηρεσία. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να δώσουμε συνέχεια και να το παρακολουθήσουμε. Επίσης συναντήσαμε τον Υφυπουργό για θέματα οικογένειας και για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Πιστεύω και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι ήταν πολύ σκεφτή. Ο Υφυπουργό μας ενημέρωσε για το Υπουργείο του και πώς εκεί εφαρμόζονται οι αρχές που διέπουν την ισότητα των φύλων μέσα από την νομοθεσία, πώς δηλαδή ε, αποκρισταλώνονται σε νόμους. Το 2009 πέρασε ο νόμος για την ε, ενδοοικογενειακή βία, μίλησε επίσης ε, για μέτρα και νομοθετήματα κατά των διακρίσεων και είπε επίσης ότι το Υπουργείο του συμμετέχει κατά 30% στην χρηματοδότηση ανέγερσης κατοικιών για γυναίκες θύματα βίας και εμπορίου γυναικών. Συμμετέχει λοιπόν στην χρηματοδότηση αυτών των έργων. Ο υφυπουργό του Υπουργείου για Ευρωπαϊκά Θέματα, ο κύριος Πλένκοβιτς, μας μίλησε για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και όλη τη διαδικασία. Αυτά λίγο πριν τα επεισόδια στο Σπλίτ στις 12 Ιουνίου. Ο υφυπουργό μας είπε ότι όλες οι δημόσιες αρχές καταδίκασαν τα επεισόδια της 12ης Ιουνίου στο Σπλίτ. Είπε ότι η Κροατία δεν συμφωνεί με καμία μορφή και δεν ανέχεται ε, καμία μορφή βίας ούτε τώρα ούτε στο μέλλον και για την ενταξιακή διαδικασία είπε ότι πάνω από χίλια νομοσχέδια έχουν εγκριθεί ή προσαρμοστεί στα πλαίσια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Την επόμενη μέρα συναντηθήκαμε με την Διευθύντρια της Κυβερνητικής Υπηρεσίας για την Ισότητα των Φύλων και την Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως και μαζί τους μιλήσαμε για τις εκάστοτε δραστηριότητες των Υπουργείων ή Υπηρεσιών τους. Η Υφυπουργός Δικαιοσύνης είναι φορτισμένη και με θέματα συνηγόρου του πολίτη και είπε λοιπόν η Υφυπουργό ότι η ατζέντα του συνηγόρου του πολίτη δεν θα αλλάξει αλλά θα ενοποιηθεί σε μια υπηρεσία. Τέλος, συναντηθήκαμε με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων και εκπροσώπους του δημοσίου τομέα. Ε, είδαμε εκπροσώπους από 10 περίπου μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αυτή η συνάντηση ήταν χρησιμότατη. Μετά από την παρουσίαση μιας μη κυβερνητικής οργανώσης, ε, ε, κάποιοι αντιπρόσωποι μετά από κάποια διαφωνία εγκατέλειψαν την αίθουσα. Εμείς ε, είπαμε ότι θα πρέπει να ε, υπάρξει συμβολή από όλους για την επίλυση των θεμάτων. Όμως υπήρξε μία ρήξη μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με διάφορους τομείς. Ε, μιλήσαμε και για τη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, μιλήσαμε για την παιδεία, τη βία, για την κατάσταση των ε, γυναικών Ρωμά στην Κροατία, για τις ε, διαφορές στους μισθούς και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των γυναικών. Τέλος, θα ήθελα να πω και να θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σβένσον που ήταν η πρόεδρος ε, και της Επιτροπής και της αντιπροσωπείας. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία και κατά την προηγούμενη και κατά τη διάρκεια αυτής της ε, θητείας του Κοινοβουλίου συμμετείχα σε πολλές αντιπροσωπείες. Αυτή η αντιπροσωπεία είχε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Είχαμε ε, αρκετό χρόνο για να προετοιμαστούμε, να κάνουμε διαπραγματεύσεις, ε, συναντήσεις με εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους όσους βοήθησαν. Και, αν μου επιτρέπετε, ε, βλέπω η κυρία Όβη δεν είναι εδώ πια. Α, ε, φαντάζομαι ότι δεν θα είχε να προσέσει πολλά πράγματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ζαμπόσκα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες ε, που μας κοινοποιήσατε σε σχέση και με την γνωμοδότηση που, την έκθεση μάλλον που έχει διανεμηθεί και είναι και στο φάκελο της συνεδρίας, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Οπότε ας περάσουμε στο επόμενο σημείο, δηλαδή εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για την ε, κατάσταση των γυναικών σε κατάσταση ένοπλη σύραξη. Η κυρία Νικολάη έχει το λόγο, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα και για να προς το για λόγους σεβασμού προς τις Ρουμάνες γυναίκες που εμπλέκονται σε διάφορες ε, σειράξεις διότι ε, η χώρα μου έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα, μεγάλο άλμα προς τα μπρος επί του θέματος αυτό. Πρέπει να ομολογήσω ότι θα προτιμούσα να μην είχα αναλάβει αυτή την έκθεση γιατί θα προτιμούσα να υπήρχε ειρήνη, να μην υπάρχουν ενόπλες σειράξεις και να μην υπάρχουν θύματα φυσικά. Αυτή είναι η επιθυμία μου, αλλά ΦΕΦ προσφάτως είχαμε αρκετές ε, καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, ε, ιδίως ε, τα όσα συνέβησαν στη Βόρεια Αφρική. Ε, πρόκειται για Συγκρούσει οι οποίες δεν ήταν μεγάλη κλίμακα, αλλά υπήρχαν και ακραία φαινόμενα βία. και φυσικά τα πρώτα θύματα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Πρόκειται λοιπόν για ένα ζήτημα το οποίο είναι επίκαιρο και απασχόλησε και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι πολλές ε, εκ των συναδέλφων γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρω ότι μετά από την ε, έγκριση του ψηφίσματος 1925 ε, του ΟΗΕ και του 1920 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη ενεπλάκει στην υιοθέτηση μέτρων προκειμένου η κατάσταση των γενικών ε, σε περιοχές όπου υπάρχουν ένοπλες σειράξεις να είναι καλύτερη. Τα κράτη-μέλη και ο ΙΕ εν γέννη στην εφαρμογή του 1325 έκανε ένα βήμα προς τα μπρος. Υπάρχει πλέον ένας ε, ειδικό εκπρόσωπος του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας ε, στη διάρκεια των έναπλων σειράξεων. Η Μάρκο του Βάλστρομ είναι αυτή. Και αυτό φυσικά αναγνωρίζει και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο ζήτημα. Επιπλέον θα ήθελα να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι θέμα της επικαιρότητα, ακόμα και αν το γεγονός ότι η πλατφόρμα του Πεκίνου συστάθηκε το 1995. Μετά από την πλατφόρμα του Πεκίνου αναλήφθηκαν μέτρα από τα κράτη-μέλη για να υπάρχουν και εθνικά μέτρα και εθνικές στρατηγικές ε, βάσει των αρχών του Πεκίνου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρεται και στο ψήφισμα του 2006 που αφορά ακριβώς το θέμα των γυναικών σε περιπτώσεις έναπλων σειράξεων, αλλά πέραν ε, της αντιμετώπισης που έχουμε σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να είναι κρίσιμη κατάσταση. Οι βασικές συστάσεις ε, της έκθεσής μου διότι θέλω να έχουμε και μία σταθερή θέση ως Επιτροπή επί του ζητήματος, είναι η εξής. Επιτρέψτε μου βέβαια πριν να αναφερθώ στην ε, κατάσταση του Συμβουλίου που έχει δημιουργηθεί τον Ιούλιο του 2010 για θέματα ασφάλειας και ειρήνης των γυναικών και ασχολήθηκε με κάποιους δείκτες που θέλουν να μελετήσουν την εφαρμογή αυτού του προγράμματος δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο κατά την άποψή μου είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα. Η σεξουαλική ε, βία μέσω μαζικών βιασμών είναι δυστυχώς κάτι το οποίο χρησιμοποιείται ακόμα ως τακτική πολέμου. Δεν εκπολιτίστηκε και πολύ η ανθρωπότητα, διότι πρόκειται για μια ε, δραστηριότητα η οποία χρησιμοποιόταν από την αρχαιότητα και εξακολουθεί να υφίσταται στον 21ο αιώνα όσοι διαπράττουν αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα δυστυχώς ε, μένουν ατιμόρυτοι, υπάρχει μεγάλο ποσοστό ατιμορρησίας, υπάρχει το κλασικό παράδειγμα της Βοσνίας υπάρχουν 13 εισαγγελείς που ασχολούνται με χιλιάδες υποθέσεις, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει σεβασμός από πλευρά κρατών μελών για το ζήτημα αυτό. Δεν θέλει να καταπολεμήσει τις συγκεκριμένε συμπεριφορές. Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες ε, στρατιώτες ε, δραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ε, αποτελούν σημείο αναφοράς σε περιοχές ενόπλης σύραξης και οι γυναίκες αυτές συνεισφέρουν στην πάταξη των ανδρικών προτύπων και στερεοτύπων που έχουν δημιουργηθεί και η βελτίωση είναι πολύ σημαντική. Παραδείγματος χάρη στο Αφγανιστάν οι γυναίκες στρατιώτες ήταν αυτές οι οποίες κατόρθωσαν να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα. Είχαμε ειρήνη στην περιοχή χάρη στη συνδρομή τους. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν περισσότερο οι γυναίκες και στην πρόληψη αλλά και στην επίλυση των σειράξεων. Γι' αυτό λοιπόν κάνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να έχουν πολύ περισσότερες γυναίκες στρατιώτες και σε υψηλές θέσεις αλλά και στις ε, βασικές ε, θέσεις ε, των ενόπλων δυνάμεων. Γυναίκες αξιωματικοί στις ενόπλες δυνάμεις είναι σημαντικό να υπάρχουν και επίσης είναι σημαντικό όχι μόνο στις στρατιωτικές αποστολές αλλά και στις πολιτικές αποστολές να είναι μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών. Διότι κατά την άποψή μου στο μέλλον η λύση των σειράξεων θα σχετίζεται και με τη σύμπραξη πολιτικού και στρατιωτικού σκέλους ε, στις περιοχές όπου υπάρχει σύραξη. Η διατήρηση της ειρήνης, οι αποστολές αποκατάσταση της ειρήνης ε, είναι ε, πολύ σημαντικές για το μέλλον και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, σημαντικό να συμμετέχουν και οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις. Αναφέρομαι σε πολιτικές, κυβερνητικές, στρατιωτικές ε, θέσεις. Η ανοχή, η διπλωματία, η δυνατότητα να υπάρχει διάλογος είναι σημαντικοί παράγοντες ε, για την επίλυση των σειράξεων σε τομείς στους οποίους ε, κυριαρχεί η βία και σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Αναφέρομαι επίσης και στην παιδεία που αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της ε, ε, συμμετοχής των γυναικών στο τομέα αυτό. Τα κράτη-μέλη έχουν κάνει πολλά επί του ζητήματος. Αλλά στον τομέα της διαμοσολεύησης θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πολύ πιο δραστήρια και θα πρέπει να εμπλέξει τις γυναίκες στις ειρηνευτικές διαδικασίες προκειμένου να συμμετέχουν και στις διεθνείς ομάδες. Δυστυχώς, από την πρόσφατη εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνουμε ότι όταν υπάρχει μία ομάδα διαπραγματεύσεων ε, η οποία αποτελείται από άνδρες, για να παραφράσω εδώ και τον Ταλερά οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν και πάρα πολύ οι γυναίκες είναι πιο αποτελεσματικές και πιο ε, συμφιλιωτικές και αυτό επιτρέπει να προχωρούν καλύτερα οι διαπραγματεύσεις. Πρόκειται για ένα χάρισμα των γυναικών και το έχουμε διαπιστώσει και ε, κατά το ρούν της ιστορίας πώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Η... Τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι θέμα πολιτισμού και τα πρότυπα τα οποία επικρατούν αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτα. Δυστυχώς όμως σε κάποιες περιοχές ε, συγκρούσεων υπάρχει ανοχή. Να μην ε, ξεχνάμε τα όσα συνέβησαν στη Ρουάντα, στην Αγγόλα και την ε, στάση της διεθνούς κοινότητας. Ήταν απλώς μια τυπική έκκληση χωρίς να υπάρξει και μεγάλη συμμετοχή. Αναφέρθηκα και στην ατιμορρησία που είχαμε σε πολλές περιοχές σύραξης σε δικαστικό επίπεδο θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην ατιμορρησία διότι η ειρήνη και η δικαιοσύνη δεν θα πρέπει να είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αναπέσπαστα μεταξύ των. Οι ε, ένοχοι λοιπόν, ανεξάρτητα από τις συνθήκες τις οποίες διαπράτεται ένα άγκλημα, θα πρέπει να ε, βρίσκονται ενώπιον των δικαστηρίων. Στην αποκατάσταση της ε, ειρήνης είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη η συμμετοχή των γυναικών. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες οι γυναίκες αποτελούν βασικό πυλώνα των κοινοτήτων αυτών και η αποκατάσταση των κοινωνιών αυτών θα πρέπει να γίνει με την υποστήριξη των γυναικών που αποτελούν και το στήριγμα της οικογένειας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προβλέπετε για την αποκατάσταση της ειρήνης μετά από συγκρούσεις ε, μια εταιρική σχέση μεταξύ κοινωνίας των πολιτών και γυναικών. Ένα βασικό στοιχείο το οποίο αναφέρω στην έκθεσή μου είναι η έκκληση που γίνεται για τη δημιουργία μια θέση ειδικού εκπροσώπου για τις ε, γυναίκες ε, στα πλαίσια της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Γιατί θεωρώ την απαραίτητη η συγκεκριμένη θέση όπως υπάρχει άλλωστε και στον ΟΗΕ, ε, ε, είπα το εκπρόσωπος. Οι σειράξεις με θύματα γυναίκες είναι πάρα πολλές πλέον και θα πρέπει να υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις ε, σε αυτή την κατάσταση. Και κατά συνέπεια απαιτείται ισότιμο επίπεδο με τον ΟΗΕ. Έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευτυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν άνδρες και γυναίκες, ε, πολιτικοί άνδρες και πολιτικές γυναίκες ή εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών που έχουν μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη επί του ζητήματος. Δεν θεωρώ ότι αποτελεί και πολύ μεγάλο οικονομικό άχθος, αλλά ακόμα και να αποτελούσε οικονομικό, ε, ε, οικονομική επιβάρευση, τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ σημαντική, διότι μέσω μακροπρόθεσμα θα είναι πολύ σημαντικές οι συνέπειες. Θα μπορέσουμε να είμαστε πιο συνεκτικοί, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το διάλογο και με τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και με τον ΝΑΤΟ επί των ζητημάτων αυτών. Θεωρώ επίσης ότι στις στρατιωτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και κάποιος ε, συμβουλευτικός ε, ρόλος ε, για τα θέματα της ισότητας των φύλων. Θα πρέπει όσοι ασχολούνται με θέματα ενόπλων σειράξεων να λάβουν υπόψη τους και τη διάσταση του φύλου. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε ε, να υπάρχουν και σύμβουλοι ειδικοί επί των ζητημάτων αυτών. αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν και εθνικά προγράμματα δράσης επί του ζητήματος λαμβάνοντας υπόψη και τα τελευταία στατιστικά δεδομένα. Υπάρχουν μόνο 10 κράτη-μέλη τα οποία έχουν συγκεκριμένες στρατηγικές επί του ζητήματος οι γυναίκες δηλαδή και η ειρήνη βάσει και του ψηφίσματος 1325. Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να συμπληρώσουν ακόμα τα προγράμματα δράσης σας. Με την άδειά σα λοιπόν δεν θα ήθελα να καταχραστώ την υπομονή σας αλλά θα ήθελα να υπενθυμισω τρει τρει-τέσσερι δείκτες. Δείκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε λίγο πώς έχει παρούσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματος χάρη, το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν στις ε, διαπραγματεύσεις ε, σε ειρηνευτικές διαδικασίες ε, τις οποίες διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2008 και τούδε είναι μόνο δύο γυναίκες οι οποίες ε, συμμετείχαν σε διαπραγματεύσεις σε χώρες όπως το Σουδάν και η Σομαλία. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία όσον αφορά το συγκεκριμένο αριθμό γυναικών που συμμετείχαν ε, στα διαδικασίες, απλώς ξέρουμε ότι δύο κράτη έστειλαν γυναίκες. Το στοιχείο αυτό βέβαια δεν θεωρείται αντικειμενικό κριτήριο, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι στο Αφγανιστάν δεν συμμετείχε ούτε μία γυναίκα. Πέντε κράτη-μέλη είπαν ότι υποστήριξαν οικονομικώς μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετείχαν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε καλύτερα και περισσότερο τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ε, οι οποίες ε, προβάλλονται καλύτερα και είναι οι πιο αποτελεσματικές στα σημεία αυτά. Επίσης, το ποσοστό των γυναικών που είχαν ηγετικούς ρόλους σε διπλωματικό επίπεδο στις 36 ε, αντιπροσωπείες υπάρχει μόνο μία γυναίκα επικεφαλής αντιπροσωπείας στην Ερυθρέα ο μέσος αριθμός γυναικών που είναι επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στα κράτη-μέλη ήταν 18%. Με την εξαίρεση της Σουηδίας όπου έχουμε ένα 34% σε ποσοστό γυναικών, ο αριθμός των γυναικών στις αποστολές του ΟΗΕ είναι μόνο 10%, η Φιλανδία όμως έχει 30% συμμετοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι βάσει και αυτών των στοιχείων καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ε, συμμετοχή γυναικών και να αποτελεί σημείο αναφοράς αυτό στις ε, ε αποστολές είτε τις στρατιωτικές είτε τις πολιτικές. Υπάρχουν και άλλα στατιστικά στοιχεία και άλλοι δείκτες τους οποίους ανέλησα. Δεν ε, θεωρώ βεβαίως ότι έχω εξαντλήσει το θέμα αυτό. Πρόκειται για ένα ευρύτατο ζήτημα, πολύ δύσκολο, αποτέλεσε πρόκληση για μένα και θα πρέπει να ομολογήσω, ειλικρινά να σας ομολογήσω, ότι για να είναι αποτελεσματική η έκθεσή μας και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση, θα πρέπει να δράσουμε και θα πρέπει να φροντίσουμε η έκθεσή μας να είναι και ε, με βάση την πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Νικολάη. Η κυρία Νάντελ Σέπα έχει το λόγο. Merci, Ευχαριστώ Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Νικολάη γιατί είναι δελεχέστατη και εξαιρετική η εργασία που έκανε για αυτό το ευαίσθητο ζήτημα. Είναι πληρέστατη η έκθεση και συμπεριλαμβάνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κατάσταση των γυναικών ε, εν καιρό πολέμου, σε ένοπλε σειράξει. Διαπιστώνουμε πόσο πολυδιάστατο είναι αυτό το θέμα και συνειδητοποιούμε ότι είναι μεγάλη η πρόκληση. Η συγγήτρια πάντως ε, κατάφερε με μαεστρία να πραγματευτεί αυτό το θέμα. Εξετάζουμε το θέμα των θυμάτων αλλά και του ρόλου που έχουν για την πρόληψη και την ε, διευθέτηση κρίσεων είτε είναι κομμάτι της σύραξης είτε είναι εκτός. Ε, νομίζω ότι σωστά τονίσατε τον κεντρικό ρόλο στις, των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις και στις επιχειρήσεις είτε είναι ένοπλες είτε όχι. Επίσης μιλήσατε για τη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσώπου δηλαδή για τις ε, γυναίκες, ε, για την ασφάλεια και την ειρήνη. Πάρα πολύ σημαντικό και σας παραπέμπω στην παράγραφο 12. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθήσει τη διαφάνεια σχετικά με τη θέση και την περάσπιση του ρόλου των γυναικών ε, ανά τον κόσμο και συμφωνώ απολύτω με τις παραγράφους 13 έως και 18 που προτείνεται καλύτερο συντονισμό τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το θέμα των γυναικών, τη ασφάλεια και τη Ειρηνή συμπερίληψη των γυναικών στι διαπραγματεύσει και στη διαχείριση διαφόρων κρίσεων και καταστάσεων, ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα προσφυλέ και υποστηρίζω από αυτού τη θέση της εισηγήτριας. Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποια ζητήματα όπου θα ήθελα να ενισχυθεί κατά τη διατύπωση. Πρώτον, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να επιμείνουμε για τι επιπτώσει τη σεξουαλική βία κατά των γυναικών και των οικογενειών του. Είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ίσω σε μια ξεχωριστή παράγραφο τι καταστροφικέ ε, συνέπειε σε σωματικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο επί των θυμάτων και επί των ε, συζύγων του ε, και των παιδιών τους ε, για όλη την οικογένεια. Δεύτερον, στην καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας θα πρέπει να τονίσουμε όπως κάνετε μέσα στην έκθεση το ρόλο των γυναικών και επίσης θα πρέπει να επιμείνουμε στις κυρώσεις, στις ένοπλες και τις παραστρατιωτικές ομάδες όταν υπάρχουν κρούσματα βίας γιατί χρησιμοποιείται η βία για να τρομοκρατηθεί ο πληθυσμό ε, και θα πρέπει να τηρείται ο εσωτερικό κανονισμό ε, βάση τη ε, εθνική νομοθεσία στον τομέα αυτό. Τρίτη διάσταση, επιμείνατε πολύ στην εκπαίδευση, στην αιτιολογική έκθεση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στο βασικό ε, κορμό του κειμένου γιατί η παιδεία, η εκπαίδευση είναι στη βάση της αλλαγής της νοοτροπίας και της αλλαγής της κοινωνίας και καλό θα ήταν να επιμείνουμε περαιτέρω σε αυτό το σημείο μέσα στην έκθεση. Τελευταίο σημείο, σεβασμός των παραδόσεων μέσα στα παιδευτικά προγράμματα, προγράμματα ευαισθητοποίησης. Στη διάσκεψη που διοργανώσαμε εδώ ε, στις 14 Ιουνίου σχετικά με την κατάσταση των γυναικών ε, σε καιρό πολέμου, μίλησα για το θέατρο, για τη ζωγραφική, για του παραδοσιακού χορού και το ρόλο που μπορούν να έχουν στα πλαίσια των προγραμμάτων ευαισθητοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα ήθελα λοιπόν να το τονίσουμε εδώ και συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν ήδη καλέ πρακτικέ και δεν αντίκειται στι παραδοσιακέ ε, και πολιτιστικέ ευαισθησίε. Μην το ξεχνάμε και αυτό, διότι πρόκειται για πολύ ευαίσθητε ε, ε, στιγμέ και νομίζω ότι είναι καλό να προαγάγουμε ήδη υφιστάμενε παραδοσιακέ πρακτικέ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια που ε, κατάφερε ε, να εκθέσει ε, με πληρότητα όλες τις διάφορες πλευρές αυτού τόσο ευαίσθητου ζητήματος. Σας ευχαριστούμε. Τώρα, εκπρόσωπο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Α, η κυρία Ζαμπόσκα. Εκπροσωπείτε την Επιτροπή, κυρία Ζαμπόσκα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να προσθέσω κάποιες παρατηρήσεις στην έκθεση της κυρίας Νικολάη. Συγχαρητήρια καταρχήν για την σύνθετη προσέγγιση αυτής της προβληματικής Ε, εκπλήσει και θορυβεί λίγο το γεγονός ότι το ψήφισμα 1325 του ΟΗΕ ε, είχε εγκριθεί πριν από 11 χρόνια. Ήδη από πριν, χρόνια πριν, η κατάσταση των γυναικών στους πολέμους σε περιοχές ένοπλων σειράξεων ήταν πολύ δυσχερής και η συγγήτριά μας είπε ότι μέσα σε αυτά τα 11 χρόνια πολύ περιορισμένη πρόοδος μόνο επιτελέστηκε και η κατάσταση των γυναικών δεν βελτιώθηκε. Αυτό μας θορυβεί και μας ανησυχεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική βία, η οποία χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου σε πολλές χώρες και ακόμη ισχύει η ατιμορρησία. Υπάρχουν πολλές γυναίκες ε, που υποφέρουν στις εμπόλεμες ζώνες για διάφορους λόγους και η συγγήτριά μας είπε ότι είναι απαραίτητο να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες σε διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. και ε, εκείνοι που μένουν σε εμπόλεμες ζώνες ισχυρίζονται ότι οι γυναίκες παίζουν ρόλο πρωτοπόρο γιατί θέλουν πρωτίστως να προστατέψουν τα παιδιά τους, την οικογένειά τους και έτσι δυσκολεύονται για τις γυναίκες αυτές ακόμη περισσότερα τα πράγματα γιατί πλήττονται καθημερινά. Μία ερώτηση κυρία εισηγήτρια να σας κάνω. Σκόπιμα ε, απαλείψατε ε, ένα στοιχείο πολύ θλιβερό το οποίο τελευταία προβάλλεται όλο και περισσότερο. Πρόκειται για τις γυναίκες τρομοκράτε, τις Δηλαδή αυτό δείχνει ότι οι γυναίκες δεν παλεύουν μόνο κατά των πολέμων στις εμπόλεμες περιοχές, αλλά υπάρχει και μια αλλαγή. Όλο και περισσότερες γυναίκες χρησιμοποιούνται ως ζωντανές βόμβες και συμμετέχουν σε τρομοκρατικά πλήγματα. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δηλαδή σε αυτό το σημείο ε, έμοιασαν μετά από κάποιο διάστημα οι γυναίκες τους άντρες και ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους και νέοι και παιδιά επίσης συχνά γίνονται τέτοιες ζωντανές βόμβες έχει να κάνει με το περιβάλλον από το οποίο προέρχονται, στο οποίο μεγάλωσαν, ε, επειδή ας πούμε προέρχονται από φτωχές περιοχές. Ίσως ε, γι' αυτό επηρεάστηκαν ή το κάνουν για να εξασφαλιστεί η οικογένειά τους οικονομικά ή οφείλεται στην απελπισία των νέων και των γυναικών που τους φέρνει να διαπράττουν τέτοιες πράξεις Ίσως δεν θα ήταν άσχημο να αφιερωθούν δύο προτάσεις στο πρόβλημα αυτό, ε, δύο παράγραφοι, ούτως ώστε να ασχοληθούμε και με το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι ένα φαινόμενο θλιβερό, που όμως πρέπει να μας απασχολήσει. Και πάλι ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για την εργασία σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσθέσω και εγώ τα, στα κολακευτικά σχόλια που έχουν ακουστεί για το σχέδιο έκθεση ότι ναι, είναι μια αξιόλογη έκθεση που έχουμε ενωπιό μα και πάντα επίκαιρη. Γιατί βλέπουμε σειράξει σε πολλέ περιοχέ, ιδίω στην Ανατολική Μεσόγειο, σήμερα στη Μέση Ανατολή και οι γυναίκε υπόκεινται σε σεξουαλική βία αλλά επιπρόσθετα θα πρέπει να τονιστεί ακριβώς και τα ψυχολογικά τραύματα που δημιουργούνται είτε στην ίδια τη γυναίκα όταν η ίδια θυματοποιείται, αλλά και στα μέλη της οικογένειας. Συνήθως αυτή η παράμετρος νομίζω δεν τονίζεται στην έκθεση. Βλέπουμε γυναίκες να βιώνουν την απώλεια συγγενικών τους προσώπων. Σε τις καθημερινέ εικόνε τη τηλεοράση μα βλέπουμε ολόκληρε οικογένειε να αφανίζονται, Οι άντρες, τα παιδιά, οι κόρε. Και έχοντα την εμπειρία και στη δική μου πατρίδα, στην Κύπρο, ακόμα σήμερα μιλούμε για τον πόνο γυναικών που ψάχνουν να βρουν αγνοούμενου. Υπάρχει το πρόβλημα των αγνωμένων μελών. Και αυτέ είναι τρομερές ε, απώλειες μέσα σε μια οικογένεια, ιδίω όταν λάβουμε υπόψη το ρόλο της γυναίκα σε μια οικογένεια. Η ίδια σαν μάνα πονή, η ίδια σαν σύζυγος από την απώλεια ή του συζύγου ή του παιδιού αλλά ειδικά στην περίπτωση αγνοωμένων είναι μια ανοιχτή πληγή. Πόσα χρόνια και να περάσουν, εάν δεν επουλωθεί με τη διακρύβωση της τύχης του αγνωμένου και με την ταφή του αγνώμενου προσώπου, πιστεύω ότι είναι μια δραματική απώλεια και τη βιώνει η γυναίκα και η, κακή της ψυχολογία μεταφέρεται και στα άλλα μέλη της οικογένειας. Επομένω, θα ήθελα στην έκθεση να μιλήσουμε λίγο και για τις απώλειες και τα ψυχολογικά τραύματα από ανοιχτές πληγές αγνωμένων μελών. Γιατί και εκεί η γυναίκα θυματοποιείται αλλά και η οικογένεια. Και επιπρόσθετα χαίρομαι γιατί τονίζεται το γεγονός ότι ένοχοι σεξουαλικής βίας χαίρουν ατιμορρησίας. Είναι γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση των δικαστών και των εισαγγελέων στην έρευνα και να τιμωρούνται ακριβώς οι βιαστές εκείνοι οι οποίοι θυματοποιούν γυναίκες, οι μέλη της οικογένειας και στις ειρηνευτικές διαδικασίες πρέπει να είναι ξεκάθαρον ότι η ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά και η δικαιοσύνη πρέπει να πονέμεται γρήγορα. Γιατί, όπως λένε οι Άγγλοι, ε, «Justice delayed is justice denied» και δυστυχώς βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι τόσο χρονοβόρες οι διαδικασίες που αν η δικαιοσύνη δεν απονέμεται και περνούν τα χρόνια τότε ακριβώς αυτή η ατιμορρησία παραμένει εκεί και δεν αποτρέπει τέτοιου είδους εγκλήματα να επαναλαμβάνονται. Επομένως θεωρώ ότι οι δύο αναφορές που γίνονται στην ανάγκη οι ένοχοι να τιμωρούνται και ότι η ατιμορρησία δεν πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμη πρέπει να ενισχυθούν και η δικαιοσύνη να απονέμεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και συμφωνώ οπωσδήποτε με την ανάγκη να δημιουργηθεί ε, ειδική θέση αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, ακριβώς για να ενισχυθεί αυτός ο τομέας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Παπαδοπούλου, η συγγητρία μας κυρία Νικολάη. Uh, Ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας. Πράγματι, όλα αυτά που είπατε είναι σημαντικά. Καταρχήν για την ψυχολογική ζημιά που υφίστανται. Σίγουρα θα αναφερθεί το θέμα αυτό στην έκθεση για δύο λόγους. Πρώτον, είναι σημαντικό σε περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο, αλλά και σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο που η βία προβάλλεται από τα ΜΜΕ παντού, αυτό γίνεται ακόμα πιο ε, σημαντικό με μέσο και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και επιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν να ε, ακολουθήσουμε μια ενωσιακή προσέγγιση προς τον ψυχολογικό αντίκτυπο και τις επιπτώσεις διότι αν το ζήτημα αυτό το αφήσουμε ε, εκτός προσοχής μας θα επιδεινωθεί και θα εντείνει τις ψυχολογικές επιπτώσεις ε, κάθε σύγκρουσης που είναι δυσμενής ούτως ή άλλως. Συμφωνώ με όλα όσα είπε η κυρία Νεντέλτσεβα, βεβαίως οι επιπτώσεις στις οικογένειες, ε, οι κυρώσεις ό,τι έχει σχέση με την παράδοση και την παιδεία πρέπει να ε, ενσωματωθεί στην έκθεση γιατί είναι σημαντικό. Ε, σύντομα για την κυρία Ζαμπόρσκα. Δεν μίλησα για τις γυναίκες καμικάζι, τις γυναίκες τρομοκράτες, γιατί είναι αυτουργοί και όχι θύματα συγκρούσεων. Η απάντησή μου εν προκειμένου είναι Θα ήθελα να απαντήσω τώρα στα γαλλικά στην ερώτησή σας. Δεν μίλησα για τις γυναίκες τρομοκράτες γιατί πιστεύω ότι είναι αυτούργοι και όχι θύματα συγκρούσεων. Πιστεύω ότι δεν είναι η φτώχεια που τις πρόχνει στις πράξεις αυτές. Μιλάμε εδώ για ένα πολιτισμικό μοντέλο ε, μέσα στο οποίο ο πόλεμος ε, θεωρείται ευθύνη των πάντων και υπόθεση όλων. Και αυτό το μοντέλο, το οποίο επηρεάζεται πολύ από τη θρησκεία, ε, προβλέπει τις ίδιες ευθύνες σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Είναι ένα θέμα να καταπολεμήσουμε αυτό το πολιτισμικό μοντέλο θα πρέπει να αλλάξουν η εκπαίδευση για παράδειγμα για να καταπολεμηθεί αυτό το μοντέλο και είναι δύσκολο να δουλέψει κανείς προς αυτή την κατεύθυνση και πάνω σε αυτό. Με ρωτήσατε επίσης πώς, πώς μπορούμε να προστατέψουμε τις οικογένειες σε περιοχές συγκρούσεων. Πολύ σωστά τα λέτε. Παράλληλα με τις γυναίκες, όλη η οικογένεια είναι ο βασικός ε, στόχος και θύμα σε αυτές τις ε, ένοπλες συγκρούσεις. Και η διεθνής κοινότητα ε, δεν απασχολήθηκε πάρα πολύ με τα προβλήματα των οικογενειών, γιατί εκεί δραστηριοποιούνται περισσότερο οι τοπικοί και εθνικοί παράγοντες. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτηκαν πώς θα βοηθήσουν τις οικογένειες, πώς θα δώσουν, αν θέλετε, μια θεραπεία και για το μετατραυματικό στρες. Αλλά αυτοί που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό δεν είναι κυβερνήσεις, αλλά μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες ε, δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές και σε αυτά τα ζητήματα. Επίσης, με ρωτήσατε για τις διαπραγματεύσεις εγώ μελέτησα το θέμα των μετασυγκρουσιακών ή μεταπολεμικών διαπραγματεύσεων. Δεν ε, είμαι ειδική σε αυτό το θέμα, αλλά το έχω μελετήσει και ξέρω πώς διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις. Ήδη από το 16ο αιώνα η αποτελεσματικότητα των διαπραγματεύσεων και η διάρκεια τους έχει κάποια εξάρτηση από την δομή ως προς το φύλλο των αντιπροσωπιών. Δηλαδή έπαιξαν πολύ θετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις οι γυναίκες στην ιστορία. Και εμείς ε, που είμαστε μητέρες ψυχολογικά αν θέλετε τίνουμε περισσότερο προς τον διάλογο, τη συμφιλίωση, τις μη συγκρουσιακές λύσεις. Αυτός ο παράγων λοιπόν πρέπει να αξιοποιηθεί στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Νικολάη. Ε, ε, Ενημέρωση τώρα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για το θέμα αυτό. Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 8η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η εξέταση των τροπολογιών 11 Οκτωβρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΔΕΒΕ ε, στις αρχές Νοεμβρίου και η ψηφοφορία στη δική μας Επιτροπή στις 21 ε, και 22 Νοεμβρίου και στη Σύνοδο του Ιανουαρίου του 2012 θα περάσει το θέμα στην Ολομέλεια. Επόμενο σημείο θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στην ε, κυρία Σινκλέρ. Είσαστε η συγγήτρια. Ευχαριστώ. Έχετε τη γνωμοδότηση μπροστά σας πριν από λίγες μέρες ε, ετοιμάστηκε. Πριν περάσω σε αυτό το θέμα της γνωμοδότησης, επανέρχομαι στην τελευταία μου παρέμβαση πριν από καμιά ώρα στην Επιτροπή και το σχόλιο που ακούστηκε εκτός μικροφώνου. Έγινε ένα σχόλιο ότι δηλαδή γιατί βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό είναι ένα επονίδι στο σχόλιο. Ο λόγος που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι εξελέγει και σε μια δημοκρατία υποτίθεται ότι προβλέπεται και η αντιπολίτευση και ότι γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων. Εγώ εκπροσωπώ μια περιοχή με 5 εκατομμύρια ανθρώπους, μεγαλύτερη περιοχή από τον πληθυσμό κάποιων κρατών μελών ολόκληρων. Μπορεί να διαφωνείτε με τις γνώμες μου, έχω όμως κάθε δικαίωμα να τις προβάλλω. Αυτή η γνωμοδότηση τώρα για την, ε, το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και την κατάσταση ε, θα βρει διαφωνούς, διαφωνούντες πολλούς συναδέλφους. Θέλω όμως να εξηγήσω το σκεπτικό της γνωμοδότησής μου αυτής. Είπα και στην Ολομέλεια και εδώ στην Επιτροπή πολλές φορές ότι είμαι κατά κάθε μορφής διακρίσεων. Η κατάσταση θα, εδώ πρέπει να αλλάξει σε όλες τις κοινωνίες θα πρέπει οι διακρίσεις λόγω ηλικίας, λόγω αναπηρίας να καταργηθεί. Όλοι είμαστε ίσοι. Προς τα εκεί τίνουμε. Αυτό θέλουμε όλοι. Όλο το θέμα όμως της κίνησης της, της ισότητας ε, είναι ότι δεν πρέπει να ε, κάνει διαφορά η ηλικία ή οτιδήποτε. Εμείς εδώ μιλάμε, είμαστε στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, όχι για πρόσθετα δικαιώματα γυναικών ή ανδρών. Μιλάμε για ισότητα. Γι' αυτό αντιτίθεμε τόσο πολύ στις θετικές διακρίσεις, γιατί οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων δημιουργεί θύματα. Και ε, το να νομοθετούμε και να δημιουργούμε θύματα έτσι, αυτό ηθικά είναι λάθος. Επίσης είμαι υπέρ των ίσων ευκαιριών ίσης μεταχείρισης για όλους. Έχουμε κάνει κάποια έρευνα που στηρίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, με παρόμοια αποτελέσματα για πολλούς. Βλέπετε εδώ στην έρευνα ότι το 86% το, του κόσμου πιστεύει ότι οποιαδήποτε μορφή προτιμησιακής ε, μεταχείρισης λόγω φύλου είναι λάθος. Είναι ενδιαφέρον να δούμε και τις επόμενες στήλε ε, που δείχνουν ότι οι περισσότερες είναι γυναίκες που πιστεύουν ότι αυτό θα ήταν λάθος. Πιο πολλές γυναίκες από ότι οι άνδρες, γιατί οι γυναίκες δεν θέλουν ε, ε να τις αντιμετωπίζουν πατερναλιστικά. Αν δούμε επίση και άλλα θέματα εκτό από το ηλικιακό, βλέπουμε ότι αυτοί που θέλουν προτιμησιακή μεταχείριση λόγω ηλικία, βλέπουμε ότι οι νέοι ως επιτοπλίστων πιστεύουν ότι είναι λίγο καλύτερο να κάνουμε κάποιες θετικές διακρίσεις από ότι οι ηλικιωμένοι. Οι ηλικιωμένοι δεν το θέλουν δηλαδή. Άρα οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι θα είναι οι δικαιούχοι των μέτρων θετικής διάκρισης είναι κατά οι περισσότεροι από αυτούς. ή στις προσλήψεις. Δεν πρέπει να παίρνουμε τον καλύτερο με βάση την απόδοση, την ικανότητα να κάνει τη δουλειά, τα προσόντα. Οι διακρίσεις τι είναι. Δεν ξέρω αν έχετε πέσει θύματα διακρίσεων. Εγώ ναι. Και είναι το πιο φρικτό πράγμα στον κόσμο. Μπείτε στη θέση ενός άνδρα για παράδειγμα που δούλεψε μια ζωή για να πάρει μια συγκεκριμένη θέση. Αυτό έγινε μάλιστα. Το Εργατικό Κόμμα είχε κάνει θετικές διακρίσεις για τις γυναίκες στο Κοινοβούλιο. Ενώ άνδρες είχαν δουλέψει χρόνια για να κατακτήσουν μια θέση και από την άλλη ο μόνος λόγος που δεν τους επετράπη να θέσουν υποψηφιότητα ήταν το φίλο τους. Αυτό δεν μπορεί παρά να είναι λάθος. Δεν μπορεί να λέμε ότι ε, μόνο και μόνο για το φύλλο ε, το οποίο έχουμε από τη γέννησή μας δεν μπορούμε να κατακτήσουμε μια θέση. Δεν, είναι να, δεν μπορούμε να λέμε ότι επειδή επί χρόνια ε, υπήρχαν διακρίσεις σε βάρος ενός φίλου, τώρα θα αντισταθμιστεί με θετικές διακρίσεις σε βάρος του άλλου. Θα πρέπει να αξίσουμε κάτω από το βερνίκι ε, αυτών των επιφανειακών μέτρων. Το, και ε, εγώ είμαι κατά των μέτρων αυτών γιατί πραγματικά είναι επιφανειακά μέτρα. Δεν εξετάζουν τη ρίζα του προβλήματος όπως καλύτερη φροντίδα για τα παιδιά, φύλαξη των παιδιών. Ε, όλο και περισσότερες γυναίκες τώρα βγαίνουν από τα πανεπιστήμια αλλά δεν κάνουν σταδιοδρομία. Γιατί συμβαίνει αυτό, αυτό πρέπει να δούμε. Φύλαξη παιδιών, εκπαιδευτικέ ευκαιρίε, αυτά πρέπει να απασχολήσουν τα κράτη-μέλη. Μπορεί δηλαδή, ανεξάρτητα από την ικανότητα μια γυναίκα να μπαίνει λόγω φύλου σε θέσει ε, με ευθύνε και να παραγωνίζονται άντρε που ίσω ε, είναι πλέον ενδεδειγμένοι. Ε, από το Ηνωμένο Βασιλείο είχαμε 16 χρόνια αρχή, πρωθυπουργό γυναίκα Μάργαρετ Θάτσερ, η Ίντιρα Γκάντι, τρία ε, ονόματα έντονων γυναικών, γυναικείων προσωπικότητων που τα κατάφεραν χωρίς κανένα θετικό μέτρο διάκρισης. Ε, ευχαριστώ πολύ, περιμένω τα σχόλιά σας με ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σινκλέρ. Η κυρία Τσεκόβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, νομοδότησή της και φυσικά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι αποφάσισε να παρακολουθάει την εφαρμογή της Χάρτης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εν γέννη. φαίνεται ότι δεν είναι απερκώς ενημερωμένο το ευρύ κοινό για το κατά πόσον ε, ε, παραβιάζονται τα δικαιώματά του. Επομένως θα πρέπει να διαβιβάσουμε σε ποια κατάσταση μπορεί κάποιος να αποτανθεί στην προστασία που προσφέρει ο χάρτης και πότε έχουμε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει πλέον να μπορούν να ζητούν βοήθεια σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται όμως από τη χάρτα και επομένως είναι εκτός δικαιοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την περίπτωση τα συνταγματικά στη, συστήματα των κρατών μελών είναι αυτά τα οποία φροντίζουν ε, τα δικαιώματά τους. Η χάρτα λοιπόν συμπληρώνει αλλά δεν υποκαθιστά τα συνταγματικά συστήματα των κρατών μελών. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή επί του θέματος και θα ήθελα να αναφέρετε κάτι τέτοιο στην πρώτη παράγραφο της γνωμοδότησης. Επίσης, συμφωνώ με τη συμπερίληψη των στοιχείων που αφορούν το πόσες γυναίκες και πόσες άνδρες ε, έκαναν ε, αναφορές ε, και πόσες απαντήσεις έλαβαν. Αυτό βρίσκεται στην πέμπτη παράγραφο, αλλά θα ήθελα να περιοριστεί μόνο στα θέματα ισότητας φύλου για την αγορά εργασίας, ιδίω όσον αφορά τις πέντε προτεραιότητες που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της του 2010 για την εφαρμογή της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτό μας προσδίδει περισσότερη διαφάνεια και μας επιτρέπει να δούμε κατά πόσον υπήρχε πρόοδος ή κάποιες αρνητικές επιπτώσεις ε, λόγω της θετικής δράσης, ε, διάκρισης που αναφέρει η γράφουσα στη δεύτερη παράγραφο. παρατήρηση όσον αφορά τα παιδιά. Τα περισσότερα στοιχεία, περισσότερες αναφορές που γίνονται και οι περισσότερες παραβιάσεις αφορούν τα δικαιώματα παιδιών. Έχουμε βάλει τα παιδιά, όπως για παράδειγμα ε, ορφανά παιδιά, παιδιά ε, τα οποία είναι θύματα εμπορίας ή ε, κοινωνικής κακοποίησης. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν τα παιδιά οι γονείς τους σε ποιον μπορούν να αποτανθούν όταν υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί κατά την άποψή μου και κατά πόσον υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών και κατά πόσον προστατεύονται τα συμφέροντά τους βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κυρία Τσεκόβα. Η κυρία Τόμσεν. Ευχαριστώ. να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση. Εγώ όμως πρέπει ταυτόχρονα να πω ότι είμαι πολύ υπέρ της θετικής, των θετικών διακρίσεων και δυσκολεύομαι να εντοπίσω τα θύματα. Η έρευνα που έγινε είναι ενδιαφέρουσα. Ξέρουμε όμως ότι ένα πρόσωπο που έχει θετική διάκριση ε, μπορεί να είναι και άνδρας. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή με την καλύτερη κάλυψη ε, των παιδιών στο Ηνωμένο, στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εδώ και 40 χρόνια έχουμε πολύ καλό σύστημα και παρόλα αυτά είμαστε στην 23η θέση όταν πρόκειται για γυναίκες σε θέσεις ιεραρχικές ε, τώρα οι γυναίκες έχουν καλύτερη εκπαίδευση από τους άνδρες, αλλά λίγες, ε, για παράδειγμα, είναι σε υψηλές θέσει στο τραπεζικό τομέα. Οι προτιμησιακές λοιπόν διακρίσεις ε, υπάρχουν και στη χώρα μου και σε άλλες χώρες. Ε, παίρνει κανείς μια θέση πολλές φορές, ε, ακριβώς επειδή είναι άνδρας και αυτό ε, μόνο με τα μέτρα θετικών διακρίσεων υπέρ των γυναικών αλλάζει. Αυτό είναι σημαντικό για τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών. Και ε, είναι θετικό το βήμα ότι ε, έχει καλυφθεί αυτό το δικαίωμα στο... από την νομοθεσία. Τώρα, για τους αναπήρους. Ε, πολλές φορές προβλέπεται η συνέντευξη. Οι, οι ανάπηροι στα κράτη-μέλη μας υπέστησαν και υφίστανται μεγάλες διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Και η δυνατότητα της συνέντευξης αποτελεί, όταν θέλουν να χτυπήσουν μια θέση, αποτελεί μια ε, κατάκτηση. Δεν πρέπει να νιώθουν θύματα λοιπόν. Επίσης σημαντικό είναι στην γνωμοδότηση αυτή να περιοριστούμε στις γυναίκες. Το θέμα αυτό αφορά τις γυναίκες. Δεν επεκτείνεται για να συμπεριλάβει τα παιδιά ή άλλες ομάδες εκτός των γυναικών. Ας μείνουμε εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τόμψεν. Η κυρία Μεντελτσέβα τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για το έργο της. Θα ήθελα να επανέλθω σε αρκετά σημεία που αναφέρονται στη γνωμοδότησή της. Καταρχάς μια πολύ γενική παρατήρηση. Κατανοώ ότι εμείς δεν έχουμε την ίδια προσέγγιση λόγω των πολιτικών μας δεσμεύσεων εκατέρωθεν, αλλά ε, θα ήθελα να υπάρχει μια πολύ πιο θετική στάση από αυτή που διαπιστώνουμε στη γνωμοδότηση που μας παρουσιάστηκε. Η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ε, πλέον έκτημα για τους πολίτες μας και Πρόκειται για θέματα τρίτης γενεάς, ε, οικονομικά δικαιώματα κλπ. βρίσκονται σε άλλη μοίρα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε περισσότερο τα στοιχεία αυτά. Καταρχάς για την αιτιολογική σκέψη α. Λέτε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να λάβουν την ερμηνεία του χάρτη όπως ε, ε, επιθυμούν ε, λάθος. Θα πρέπει να ενσωματώσουν την ε, ε, ε, θεμελιώδη δικαιώματα στη χάρτα τους. Θα πρέπει να δεχτούν τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και το δικαστήριο προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και βάσει το ευρωπαϊκό δικαίωμα και θα πρέπει να γίνει βάσει της ε, συγκεκριμένης ε, παράδοσης ε, που υπάρχει σε κάθε κράτος μέλος. Εδώ έχουμε το σύνδεσμο μεταξύ συνταγματικού δικαίου μιας χώρας και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να γίνει σεβασμός του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά δεν θα πρέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο να σέβεται κάθε κράτος μέλος και κάθε συνταγματικό σύστημα κράτους μέλους. Όσον αφορά τις θετικές διακρίσεις, ναι, σαφώς μπορεί να υπάρξουν και θύματα, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει μια τέτοια δήλωση συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Η θετική διάκριση είναι ένα αγκαίο μέτρο, ε, το οποίο κάποιες φορές πρέπει να είναι προσωρισμό Μπορεί να ζητούμε, για παράδειγμα, ισότητα μισθών, στα, η συμμετοχή των γυναικών στα δυτικά συμβούλια επιχειρήσεων και αυτό δεν δημιουργεί θύματα, απλώς είναι κοινή λογική. Για την αιτιολογική σκέψη 3, λέτε ότι θα πρέπει να σεβόμαστε πλήρως ε, τον εθνική ε, παράδοση, και την ποικιλομορφία. Δεν τίθεται θέμα πολιτισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εθνικό επίπεδο. Στη χώρα μου ε, νομίζω ότι υπάρχει ένας πολιτισμός και νομίζω ότι αυτό είναι το ίδιο και για όλα τα κράτη-μέλη. Ε, είναι ε, κοντόφθαλμος τρόπος αντιμετώπισης των ζωμάτων αυτών και δεν ε, λαμβάνει υπόψη του επαρκώς την ποικιλομορφία. Στην αιτιολογική σκέψη 6 είμαι απόλυτα αντίθετα. Πώς μπορούμε να αποτελούμε, ε, να απαιτούμε να γίνεται εξέταση πρώτης ένταξης και να ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αναστολή όταν θεωρούμε ότι υπάρχει παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, το 2004 και το 2007 υπήρχε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε δύο κατηγορίες κρατών μελών. Και πώς μπορούμε να ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και αναδρομικά το ζήτημα από το 2004. Το 1973 το Ηνωμένο Βασίλειο εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαμε να τα εξετάσουμε και από εκεί. Θα πρέπει να δούμε όλα τα κριτήρια ένταξης και δεν είναι δυνατόν να επανέλθουμε σε όλα τα κριτήρια ένταξης. Θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της εφαρμογής της χάρτας σε όλα τα κράτη-μέλη και εγώ είμαι αντίθετη στην δημιουργία ενός μηχανισμού καταρχάς πώς θα δικαιολογηθεί και πώς θα δούμε την εφαρμογή και σε ποια κράτη-μέλη θα μπορούσαμε να το επιβάλλουμε υπό την ε, ε, δικαιολογία ότι είναι τα τελευταία κράτη-μέλη που εντάχθηκαν. Θα θεωρούμε ότι έχουμε πολύ της δευτέρας κατηγορίας και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ναντελσέβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Παπαδοπούλου ευχαριστώ Είμαι σκιώδης εισηγήτρια εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και ε, διάβασα επαγγελμένα αυτές τις έξι παραγράφους, αλλά ομολογώ να πω ότι το γενικότερο πνεύμα είναι ε, ε, σφαλμένο, διότι υποτιμά την ζωτική σημασία της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της προστασίας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας ακούσει την κυρία Σιγκλέρ την εισηγήτρια, θα πρέπει να αναφερθώ στα εξή. Ε, ναι, είναι τρομερή η διακριτική μεταχείριση. Ναι, ε, θέλουμε να μεριμνήσουμε ώστε ε, να ε, κατοχυρωθεί η ισότητα των δύο φύλων και να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση, είτε μιλάμε για άντρα είτε μιλάμε για γυναίκα. Ε, ναι, υπάρχουν νέε μορφέ διακριτική μεταχείριση. Όμω αυτή η έκθεση δεν έχει ω αντικείμενο την θετική ε, διακριτική μεταχείριση ούτε και τι νέε μορφέ διακρίσεων. Η συγγετρία θα πρέπει να διευκρινίσει πληθώρα ζητημάτων που αναφέρω σε αυτέ τι έξι παραγράφου. Α πάρουμε την πρώτη παράγραφο όχι, ας πάρουμε την αρχή. Ε, διαφωνούμε με αυτήν την ερμηνεία της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τα θεμελιώδη δικαιώματα αναφέρονται ρητά και με σαφήνεια σε αυτή τη χάρτα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ε, περιθώριο για παρανόηση. Αν διαβάσετε το προήμιο της χάρτα, σαφέστατα ότι η χάρτα επιβεβαιώνει ποια είναι ε, τα καθήκοντα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την αρχή της, ε, αρχή της επικουρικότητας όπως πηγάζει από τις συνταγματικές παραδόσεις και ε, τις διεθνείς υποχρεώσεις που είναι κοινέ για όλα τα κράτη-μέλη ως εκ τούτου. Η χάρτα δεν θεσπίζει καμία νέα εξουσία, κανένα νέο καθήκον για την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε τροποποιεί τι εξουσίε και αρμοδιότητε όπω ορίζονται από τι συνθήκε. Αν η εισηγήτρια θέλει να κάνει κάτι παραπάνω και να γύρει παραδείγματο χάρη ζητήματα σε σχέση με την άσκηση τη θετική ε, διάκριση ή για νέε μορφέ ε, ε, διακριτική μεταχείρηση. Αυτό υπερβαίνει το στόχο τη ίδια τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων και είναι πλήρη με λύση η για νεε διότι διακριτικη μεταχειρισης μπορούμε σε έκθεση τη ιδια τη χαρτα θεμελιωδων δικαιωματων και ειναι πλημελη η προσεγγιση διοτι δεν μπορουμε σε εκθεση τη επιτροπη μα που πραγματεύεται την ισότητα των δύο φύλων να θέσουμε λοιπόν νέα θέματα γιατί υπερβαίνουμε έτσι το πεδίο δραστηριοτήτων της Επιτροπής μας. Η συγκήτρια επίση πρέπει να εξηγήσει και να διευκρινίσει τι εννοεί όταν μιλάμε ε, για την, ε, τα θύματα τη θετική ε, διακριτική μεταχείριση. Ποια είναι αυτά τα θέματα, θα, θύματα, θα πρέπει να το προσδιορίσει επακριβέστερα, γιατί υπάρχουν πολλέ κλισέ, πολλέ γυναίκε που τη σήμερα ημέρα έχουν ε, καλύτερες επαγγελματικές δεξιότητες, μεγαλύτερη εμπειρία και παρόλα αυτά δεν μπορούν ε, να βρουν κάποια θέση απασχόλησης. Αν ε, προσωρινά χρησιμοποιήσει κάποιο τη θετική διακριτική μεταχείριση, δίνει σε αυτές τις γυναίκες τη δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Λοιπόν, η θετική διάκριση δεν είναι ένα μέτρο που αποσκοπεί στη διεύρυνση της διακριτικής μεταχείρισης. Είναι ένα μέτρο που αποσκοπεί ε, στην ε, υποστήριξη ε, του θύματος της διακριτικής μεταχείρισης για να εισέλθει στην αγορά εργασίας ή για να έχει κάποια άλλη ευκαιρία που ο δεν θα είχε. Θα πρέπει επίσης η συγγήτρια να διευκρινίσει κάποιες άλλες προτάσεις, φρασιολογίες που χρησιμοποιεί ε, ε, ευάλωτες ε, ομάδες, υφιστάμενα χάσματα, existing gaps λέει στα αγγλικά. Σε όλες τις παραγράφους η διατύπωση πρέπει να διευκρινιστεί και καλυμμένη ουδετερότητα. Τι εννοεί όλες αυτές οι διαφορές στις οποίες αναφέρεστε δεν, είναι, δεν εκφράζονται με σαφήνεια και κυρίως παρακαλώ να προσδιορίσετε ποια είναι τα θύματα εδώ γιατί μιλάμε για δύο φύλλα τις γυναίκε και τους άντρε. και συχνά λέμε στην Επιτροπή μας ότι οι γυναίκες υποφέρουν λόγω των κλισέ, λόγω της ε, διακριτικής μεταχείρισης. Λοιπόν, όπως έλεγα, είμαστε κατά των στερεοτύπων και ε, δυσκολευόμαστε εδώ να καταλάβουμε για ποια θύματα μιλάτε. Χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για την μεταχείριση επί τη βάση φύλου Επίσης οι καταγγελίες πόσες γυναίκες ε, και πόσοι άντρες ε, ε, απέστειλαν επιστολές, καταγγελίες, αναφορές κτλ. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ποιοτική διάσταση, όχι η ποσοτική. Οι ποιοτικέ αναφορές. Ποιοι είναι αυτοί που υπέβαλαν αναφορές και για ποιου είδους μεταχείριση. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε και τέλος στην τελευταία παράγραφο μιλάμε για τα παλιά και για τα νέα μέλη. Επιστέψαμε και αυτό ε, χρήζει διευκρίνηση. Ε, ε, μιλάτε εδώ για εκκρεμεί δεσμεύσει. Ποιε είναι αυτέ και ποια κράτη-μέλη δεν έχουν ε, συμμορφωθεί ε, σε αυτές τις απαιτήσεις Δηλαδή τι, τα παλιά κράτη-μέλη ε, συμμορφώνονται με αυτές τις ε, ρήτρες ενώ τα νέα κράτη-μέλη όχι. Υπάρχει σύγχυση. Επίσης δεν πρέπει να κατονομάζουμε ένα κράτος μέλος ή μια ομάδα κρατών μελών κατά αυτόν τον τρόπο, διότι το αντικειμενικό μας συμφέρον είναι η συνολική και καθολική εφαρμογή ε, ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επίσης να αναφέρουμε τα πορίσματα του Ινστιτούτου για την ισότητα των δύο φύλων και σε περίπτωση παραβιάσεων των δικαιωμάτων πρέπει πολύ συγκεκριμένα με μεγάλη σαφήνεια να αναφέρεται στα περιστατικά η συγγήτρια αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να δεχθούμε το περιεχόμενο της έκθεσής της. Επίσης πιστεύω πως θα ήταν καλύτερο να αναδιατυπώσει την έκθεσή της και ε, εφόσον με τους ε, υπόλοιπους σκιώδεις από το ΕΛΚΑ και από τους Πράσινους είχαμε ένα προσχέδιο, ήταν εκεί ε, όταν έγινε η πρώτη συζήτηση αλλά δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε το σχέδιο διότι έλειπε η συγγήτρια Οπότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε κατά τη γνώμη μας το πνεύμα της έκθεσης. Ε, αν δεν έχουμε μια έκθεση που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία, ε, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε μόνο με τροπολογίες, γιατί οι τροπολογίες δεν θα αλλάξουν το πνεύμα, τη φιλοσοφία του κειμένου. Σας ευχαριστούμε ε, κυρία Παπαδοπούλη. Κυρία Έκ έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την εργασία που διαχετεύτηκε εδώ στην έκθεση, στην ομοδότηση και εγώ έχω κάποια ερωτηματικά και σχόλια επί του κειμένου. Καταρχήν, είτε μιλάμε για τη σύμβαση, μιλάμε, είτε μιλάμε για τη σύμβαση του ΟΗΕ ή για τα βασικά νομικά μέσα της Ένωσης, πρόκειται για νομικά κείμενα που υπεγράφησαν από τα κράτη-μέλη. Άρα τα κράτη-μέλη νομικά είναι αναγκασμένα να εκπληρώσουν τον κανονισμό. Γι' αυτό γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση για την επικύρωση διεθνών ε, κειμένων. Ο χάρτης εξετάστηκε, για παράδειγμα, και από το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο επ' αυτού του θέματος. Υπάρχει μια θεμελιώδης παρανόηση σχετικά με την ιεραρχία των ε, νομικών κειμένων στην αρχή της γνωμοδότησης. Η ομάδα μας των φιλελευθέρων θα υποβάλει μια σειρά τροπολογιών για να διορθωθεί το σημείο αυτό. Δεύτερον, νομίζω ότι ακολουθούν κι άλλες παρανοήσεις και σοβαρότατες διαφορές μεταξύ των μεταφράσεων. Σουηδικά, αγγλικά, γαλλικά για παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν και γλωσσικά να εξετάσουμε το κείμενο, ίσως λόγω αυτής της ασάφειας που υπάρχει ή της θολής γνώσης σχετικά με την πραγματικότητα ε, εις ό,τι αφορά τη νομική κατάσταση. Επίσης, ε, η άποψη για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι εσφαλμένη Βεβαίως τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεργάζονται με εκπροσώπους της κοινωνία των πολιτών και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά είναι ελεύθερες και να εργαστούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις χωρίς τις κυβερνήσεις, με βάση τις δικές τους προϋποθέσεις, τουλάχιστον σε δημοκρατικά κράτη. Τώρα για την θετική, τις θετικές διακρίσεις, αυτό το σχολίασαν πολλές συνάδελφοι και συμφωνώ μαζί τους και με την άποψη της κυρίας Παπαδοπούλου συμφωνώ επί του προκειμένου, οπότε δεν πάω εγώ παραπάνω να προσθέσω. Επίσης υπάρχει μία ε, αναφορά σε σχέση με την ετήσια συζήτηση για την κατάσταση για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αν ε, δεν νομίζω ότι έχει σημασία αν απευθύνει κάποιος μια επιστολή ως άνδρας ή γυναίκα. Το περιεχόμενο μετράει και το περιεχόμενο εξετάζεται στην ετήσια έκθεση. Οπότε υπάρχει και ένας κυκλικός τρόπος, αν θέλετε, επιχειρηματολογία στην παράγραφο 5. Τα... Άρα τα επιχειρήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 6 δεν χρειάζονται, διότι η ετήσια έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων λαμβάνουν υπόψη ε, το αν κάποιο κράτος μέλος, είτε βόρειο, είτε νότιο, είτε ανατολικό, είτε δυτικό, πληρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, Επίση δεν συμφωνούμε να απομονωθούν κάποια κράτη-μέλη και τα καινούρια ε, εμπροκειμένο, γιατί δεν είναι άγια τα παλιά ε, στο συγκεκριμένο θέμα. Δείτε και την ομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να το ε, βεβαιώσετε αυτό. Και στη Σουηδία υπάρχουν, ε, για τη, Σουηδία υπάρχουν αποφάσεις του δικαστηρίου που βεβαιώνουν ότι παραβίασε η Σουηδία τη νομοθεσία για αυτά τα θέματα. Αυτά συμβαίνουν σε όλα τα κρατη Και για να κλείσω, υπάρχουν, υπάρχει ένας αριθμός μη ορθών ισχυρισμών. Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις ε, και υπάρχει μία έτσι επιχειρηματολογία όχι πλήρης και η ομάδα των φιλελευθέρων θα υποβάλει τροπολογίες για να διορθώσει τα πράγματα. Ευχαριστούμε η κυρία Βέρτμαν τώρα. Ευχαριστώ. Πολλά ακούσαμε, με πολλά συμφωνώ και εγώ. Θέλω να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, τι σημαίνει θετική διάκριση. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει γυναίκα μια θέση επειδή είναι γυναίκα και μόνο, αλλά θα έχει τις ίδιες προϋποθέσεις με τον άντρα, τα ίδια προσόντα, μόνο τότε. Και μπορεί τότε να προτιμηθεί η γυναίκα, σε εισαγωγικά το λέω αυτό. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να παρατηρήσω στη συζήτηση είναι ότι θα ήθελα μια διεξοδική εξήγηση της παραγράφου 4 που είναι πολύ ασαφής ή πρέπει να διαγραφεί ή θα πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά που αποσκοπεί. Και εμείς θα υποβάλλουμε τροπολογίες βέβαια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι η γνωμοδότηση αυτή θα έδινε το έναυσμα για τόσο μεγάλη συζήτηση. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Καμιά διάκριση. Ούτε οι θετικές διακρίσεις κάνουν καλό τα συνταγματικά δικαστήρια και οι δικαστές των συνταγματικών δικαστηρίων σε όλες τις χώρες θα ταχθούν κατά ασδήποτε μορφής διακρίσεων. Οπότε εγώ βλέπω ένα πρόβλημα εδώ. Δηλαδή, πώς θα ορίσουμε, ας πούμε, τις ε, θετικές διακρίσεις. Πίσω από αυτές τις λέξεις ε, ε, κρύβονται διαφορετικά νοήματα και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ θετικών διακρίσεων και ε, θέσεις ορισμένων όρων και προϋποθέσεων για ευάλωτες ομάδες που χρειάζονται κάποια υποστήριξη. Αυτό δεν είναι θετική διάκριση. Θετική διάκριση γίνεται όταν κάποιος ε, πάρει κάτι που δεν καλύπτεται από τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα. Εγώ είμαι κατά ιασδήποτε μορφής ε, διακρίσεων και των θετικών. Επίσης κάτι άλλο που θέλει να πει η κυρία Σίνκλερ, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, αλλά στην παράγραφο α της γνωμοδότησης ε, λέγεται ότι οι δικαστικές αρχές των κρατών μελών είναι ανεξάρτητες στην δική τους ερμηνεία του χάρτη. Αυτό σίγουρα δεν ε, συνάδει με, το, με την παράγραφο 6. Αν θέλουμε να τηρήσουμε το α, δεν μπορούμε να τηρήσουμε το 6. Και αντίστροφα, δεν ε, ταιριάζουν αυτά τα δύο. Υπάρχει ένα λάθος εδώ. Εγώ σαφώς είμαι κατά της δημιουργίας δύο κατηγοριών κρατών μελών παλαιών και καινούριων σε σχέση με την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Σινκλέρ ότι ε, η εθνική και πολιτισμική διαφορετικότητα των εθνικών κρατών πρέπει να γίνεται σεβαστή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε η κυρία Φιγκυρέιντο τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω και εγώ διάφορους ενδιασμούς. για το σχέδιο έκθεσης. Αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω εγώ, θα είμαι σύντομη. Ε, για τα συγκεκριμένα μέτρα του σημείου 2. Ε, νομίζω ότι εδώ ε, θα πρέπει να διευκρινιστεί κατά το δέον τι εννοούμε δηλαδή με αυτή την έννοια της θετικής διακριτικής μεταχείρισης, τι εννοούμε με αυτά τα θετικά μέτρα που πρέπει να αναλυφθούν για να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες η παράγραφος αυτή πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να διευκρινιστεί. Επίσης, σε σχέση με το σημείο 4, υπάρχουν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την έννοια της ουδετερότητας και ε, με την ε, σημασία που έχει η ουδετερότητα κατά την εφαρμογή της. Επίσης, συμφωνώ ότι είναι περίπλοκο πολύ το κείμενο στο σημείο 6 και γίνεται αυτή ε, η διχοτόμηση ε, ανάμεσα ε, στις χώρες, τις παλιές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις νέο αφιχθήσεις, ας τις πούμε έτσι, χώρες. Ε, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί το θέμα για να μην ερμηνευθεί, παρερμηνευθεί η διατύπωση ως διάκριση ανάμεσα στα παλιά και τα νέα κράτη-μέλη. Ε, προσυπογράφω και τις υπόλοιπες παρατηρήσεις των συναδέλφων. Εν κατακλεί, θα έλεγα ότι χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά. Ε, πρέπει να βελτιωθεί το σχεδίο για να μην ακολουθήσει οι κατευθύνσεις που είναι άγνωστες στην πορεία της Επιτροπής μας. Ευχαριστούμε κυρία Φιγκυρέιντο. Τώρα... Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Τρυς. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση για την εφαρμογή της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα λάβει υπόψη όλες τις συστάσεις σας, ιδίως κατά την εκπόνηση της έκθεσης του 2011, η οποία είναι καθοδόν. Όπως γνωρίζετε, ένας από τους στόχους ε, της έκθεσης για την εφαρμογή της ε, Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ήταν να ξεκινήσει μια ετήσια συζήτηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων και χαίρομαι ε, διότι μπορώ να σας αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ήδη τα συμπεράσματά της πριν από κάποιους μήνες. Ένας ακόμα στόχος της έκθεσης είναι να κάνει μια καταγραφή της εφαρμογής ε, της χάρτας σε όλο το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν καλύπτονται μεν όλα τα δικαιώματα, αλλά έχουμε αρκετά στοιχεία για να σας παρουσιάσουμε ε, το το περιεχόμενο των αναφορών ε, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα τα δείτε στο σύντομο αυτό φυλάδιο ε, βιβλιαράκι το οποίο εξ όσων καταλαβαίνω έχετε ήδη λάβει. Αν δεν το έχετε ήδη λάβει θα το λάβετε εντός των επόμενων εβδομάδων στη γλώσσα σας και θα είναι διαθέσιμο φυσικά και στην αγγλική γλώσσα εάν το επιθυμείτε. Ένας εκ των στόχων της έκθεσης είναι επίσης να μας δώσουν και πληροφορίες για το πού ισχύει η χάρτα. Μία από τις διαπιστώσεις μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει αρκετές επιστολές, τις οποίες ο πολίτης δεν γνωρίζει σε ποιον θα πρέπει να αποτανθεί σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών του δικαιωμάτων και γι' αυτό θα πρέπει να ενημερώσουμε καλύτερα τους πολίτες πού ισχύει ο χάρτης, σε ποιε περιπτώσεις, διότι δεν ισχύει σε όλε τις περιπτώσεις, ισχύει μόνο στις περιπτώσεις τις οποίες τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ευρωπαϊκό δίκαιο. Ισχύει φυσικά και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε μέσω παραδειγμάτων πού ισχύει η, χάρτα και πού δεν ισχύει για να μπορούν οι πολίτες να αναγνώσουν με εύκολο τρόπο, ελπίζω, ε, πότε ισχύει ο χάρτης, σε ποια περίπτωση. Να σας πω επίσης ότι θα μελετήσουμε τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όσο σας, όπως σας είπα θα τα εισλάβουμε και υπόψη ε, κατά την ε, προετοιμασία της επόμενης έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Σίνκλερ, η συγγετρία θα πάρει πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ζωντανή και έντονη συζήτηση και αντίδραση. Ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις τους. Το πρώτο που θέλω να διευκρινίσω είναι η παράγραφος 6 ε, ζητώ συγγνώμη αν ε, η ερμηνεία είναι ότι θέλω να δημιουργήσω δύο κατηγορίες ή δύο επίπεδα ή θέλω να κάνω διακρίσεις σε βάρος κάποιων κρατών μελών. Ε, τίποτα πιο μακριά από τη σκέψη μου. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα έπρεπε να ανασκευάσουμε λίγο την κατάσταση. Όταν ε, έγιναν οι προσχωρήσεις οι τελευταίες, το τελευταίο κύμα, δόθηκαν πολλές υποσχέσεις σε σχέση με το πώς θα ανέβαζαν τον πύχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι προφανές ότι πολλές χώρες δεν το έκαναν αυτό. Αυτό ήθελα να πω πριν προχωρήσουμε στα στο δεύτερο επίπεδο, ας δούμε τι έγινε με τις προηγούμενες υποσχέσεις για να δούμε και που οδεύουμε. Για παράδειγμα, ε, οι διακρίσεις ε, για τον γενετήσιο προσανατολισμό. Οι ανατολικές χώρες ε, εδώ δεν έχουν καθόλου καλά αποτελέσματα. Κανείς δεν το αρνείται αυτό. Και όμως έδωσαν συγκεκριμένες υποσχέσεις όταν έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και 7 χρόνια αργότερα που το συζητάμε το θέμα βλέπουμε ότι δεν σημειώθηκε καμία αλλαγή. Αυτό εννοώ. Πριν πάμε ένα βήμα παραπέρα, ας δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω είναι για τις επιστολές. Βεβαίως δεν μιλάμε μόνο για τους αριθμούς και θα πρέπει να δείξουμε και κάθε φορά ποιοι ήταν οι συγκεκριμένοι πέρα από τους αριθμούς για να δούμε και τι απασχολεί τον κόσμο. Νομίζω η κυρία Ντελτσεβα, συγγνώμη που δεν την προφέρω καλά, είπε ότι υπερισχύει το ενωσιακό δίκαιο του εθνικού νόμου. Ε, συγγνώμη, αλλά σε κάθε μορφή κυβέρνησης θα πρέπει να κυβερνάει η βούληση των πολιτών. Και τέτοιες έρευνες αυτή η επιστημονική έρευνα που έγινε για ε, δημοσκόπηση και έχει περιθώριο σφάλματος μόνο 3%. Όταν βλέπουμε ότι 86% του κόσμου να λένε ότι κάνετε λάθος ε, και εσύ δεν το ακούς αυτό, εμείς δεν το ακούμε, ε, θα πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν οι πολίτες. Ε. Και ε, δείτε τις γυναίκες, δείτε τα στοιχεία και τις γυναίκες. Περισσότερες γυναίκες είναι αυτές που αντιτίθενται στις θετικές διακρίσεις. Πιο πολλές γυναίκες από ότι άνδρες. Ε, εγώ εκπήρας ακούγοντας τους ε, ψηφοφόρους μου λένε ότι δεν θέλουν να τους πατρονάρουν και λένε ότι οι ποσοστώσεις δεν είναι καλό πράγμα. Εντάξει, σέβομαι τη γνώμη σας που λέτε ότι είναι καλές οι ποσοστώσεις, αλλά υπάρχει και άλλη άποψη και πρέπει να υπάρχει και μια διαφορετικότητα, μια ποικιλομορφία μεταξύ κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, εγώ καταλαβαίνω τι θέλετε να κάνετε και δεν συμφωνώ, αλλά σίγουρα πρέπει να δεχτούμε ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί. Έχουμε διαφορετικές αξίες. Ακόμα και μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν διαφορετικές ε, αξίες ε, μεταξύ Αγγλίας, Ουαλίας, Σκοτίας, Βόρειας Ιρλανδίας παρόλο που συμβιώσαμε 4-5 αιώνε και δεχόμενοι τις διαφορές ή όχι. Δεν μπορούμε λοιπόν μέσα σε 20 χρόνια να ε, απαλείψουμε ε, βασικά χαρακτηριστικά εθνικών πολιτισμών. Δεν γίνεται αυτό. Επίσης κάτι άλλο που είπε η κυρία Νεντέλτσεβα Ε, που ζητούμε ίση εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Και εγώ θα το έλεγα αυτό. Είμαι υπέρ της ίσης εκπροσώπησης, αλλά ο εξαναγκασμός από το δικαστικό σύστημα δεν είναι καλό πράγμα. Και όπως είπε και η κυρία Ζαμπόρσκα, όταν πάει στη δικαστική εξουσία ένα θέμα πολλών κρατών μελών, η ε, φυσική δικαιοσύνη προλαμβάνει τις διακρίσεις. Θέλω να πω ότι όταν ε, αναλαμβάνεται κάποια δράση και σίγουρα ε, άμα αναλυφθεί η δράση θα καταλήξουμε να ε, δούμε έναν άντρα... Παρ' όλα αυτά, οι θετικέ διακρίσει σε τελευταία ανάλυση ε, βλάπτουν τι γυναίκε. Μπορούμε να δούμε εδώ και την απόφαση του δικαστηρίου για τι ασφάλειε των αυτοκινήτων. Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα είναι πολύ πιο δύσκολο να συνδυάζεται η οικογενειακή και η επαγγελματική ζωή. Πολλέ φορέ οι θετικέ διακρίσει γίνονται μπούμεραν σε βάρο των γυναικών. Εγώ θα, με ενδιαφέρον θα συνεργαστώ με τις σκιώδεις εισηγήτριες Α, θα ήθελα να πω κάτι για τις Σκιώδης. Απογοητεύομαι λίγο γιατί η δεύτερη σε μέγεθος ε, ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι σοσιαλιστές ε, επέλεξαν αναπληρωματικό και όχι τακτικό μέλος για σκιώδη συγγήτρια. Σας ευχαριστούμε κυρία Σινκλέρ. Εκτάκτως θα ακούσουμε και την κυρία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ. Έχω μία πρόταση Διαδικαστικό είναι μάλλον το θέμα. Κάποιος που έχει μεγάλη εμπειρία με τις εμπειρολογικές και συσσολογικές έρευνες, εγώ δηλαδή, θα μπορούσε να προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσουμε διάφορες εκθέσεις που έχει στην κατοχή της η Επιτροπή. Ε, ε, αν αν βασιστούμε στις εκθέσεις που έχει η Επιτροπή μας, ε, μπορεί ε, να κλείνουμε υπέρ μιας ε, μια θέση εσφαλμένα. μπορεί κάποιο να ισχυριστεί ότι κάτι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ενώ δεν ισχύει αυτό. Μα τι σημαίνει η θετική διάκριση. Όποιος ακούει την ε, λέξη διάκριση αντιδρά τις περισσότερες ε, φορές αρνητικά. Οπότε ε, γιατί ξαφνιάζεται με το 60% η κυρία Σινκλέρ. Μπορεί κάποιος να ερμηνεύσει πολύ διαφορετικά την έννοια της θετικής διάκρισης. Εντελώς διαφορετικά από τη δική μας ερμηνεία. Οπότε αν υπάρχει μια τέτοια έκθεση, προτείνω η Γραμματεία να εξετάσει αυτή την έκθεση και αν η έκθεση βασίζεται όντως στην έρευνα και είναι εμπεριστατωμένη, καλό θα ήταν να ε, προτινόταν τότε στην Επιτροπή μας, αλλιώς ε, δημιουργούνται έτσι πλημελείς ιδέες. Σας ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε τώρα και την κυρία Σινκλέρ. Ευχαριστώ να κάνω και ένα σχόλιο σχετικό. Είπε η συνάδελφος ότι ε, είναι ειδικό σε αυτό το τομέα και ε, ε, είπε ότι είναι εντελώ λανθασμένα τα ερωτήματα. Μα εδώ είναι Δείτε ε, στη σελίδα 3, στον πίνακα 2, δεν μιλάμε για τη θετική διάκριση. Η ερώτηση είναι, πιστεύετε ότι είναι ε, αποδεκτό ή όχι να ε, χρησιμοποιεί κάποιος διακριτική μεταχείριση για να καταλάβει μια θέση εργασίας. Αυτή ήταν η ερώτηση που θέσαμε στις γυναίκες. Δεν μίλησε κανείς για θετική διάκριση. Αυτό είναι και είναι μια ανεξάρτητη ε, εταιρεία δημοσκοπήσεων έτσι, που έκανε τις ερωτήσεις. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ε, η κυρία Ιστρέλα, ευχαριστούμε κυρία Σινκλέρ. Θα κάνω ένα σχόλιο μόνο για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στην κυρία Παρβάνοβα και την κυρία Σινκλέρ. Οι μελέτες χρησιμοποιήθηκαν ως έρισμα, αλλά δεν αναφέρονται καν μέσα στο σχέδιο έκθεσης. Ε, σε κάθε περίπτωση θα έχουμε την ε, ε, ευκαιρία να επανέλθουμε στη συζήτηση αυτής της έκθεσης και να αποτιμήσουμε και πάλι ε, το περιεχόμενο των τροπολογιών. Να σας πω και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε για τις τροπολογίες 5 Οκτωβρίου μέχρι το μεσημέρι, Σεπτεμβρίου συγγνώμη, 12 το μεσημέρι και όπως αποφασίσαμε στην τελευταία συνεδρία θα εξεταστούν τροπολογίες. Ε, η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου ε, και ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ 17 Οκτωβρίου που είναι και καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Επόμενο σημείο εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης για την υποστήριξη προς το ποινικό, ε, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που υπάρχουν ε, και ο κύριος Σιμάνσκι είναι ο εισηγητής μας. Παρακαλώ. Κυρίε και κύριοι, σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης για την υποστήριξη ε, Τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ το διεθνέ Παιδικό Δικαστήριο ασχολούμαστε με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα Πρόκειται για όσους έχουν διαπράξει πολύ σοβαρά εγκλήματα κατά γυναικών και παιδιών σε μαζική κλίμακα και σε ένοπλες σειράξεις. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την προσαγωγή εγκληματιών πολέμου. Άρχισε τις εργασίες του γύρω στο 2000 και υπάρχουν πολλές ε, δίκες εν εξελίξη. Φέτος ε, το δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα ε, σύλληψης για το Μαμάρ Καντάφη και σχεδόν τη μισή υπηρεσία πληροφοριών της Λιβύης κατηγορούνται για μαζικά εγκλήματα κατά των γυναικών, για εκφοβισμό πολιτών. Αλλά δυστυχώς η αποτελεσματικότητα του δικαστηρίου περιορίζεται λόγω έλλειψης αλληλεγγύης σε διεθνές επίπεδο. Το Ισραήλ, για παράδειγμα, δεν έχει κυρώσει την ε, ιδρυτική ε, σύμβαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και η Ρωσία ή η Κίνα δεν προσχώρησαν ποτέ. και κάποια μέλη του ποινικού δικαστηρίου δεν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του. Λόγω λοιπόν έλλειψης αλληλεγγύης και λόγω και του γεγονότος ότι κατά κάποιο τρόπο το δικαστήριο είναι απομονωμένο, χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αναλάβουμε τα ενία στο διεθνές προσκήνιο και να επιβάλλουμε κάποιους όρους ε, για τη βοήθεια που παρέχεται σε τρίτες χώρες, η οποία θα παρέχεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσουν στις συνθήκες του ποινικού δικαστηρίου. θα πρέπει επίσης να αναλάβουμε και απαραίτητη δράση προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους διπλωματικούς μας να προσχωρήσουν ε, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συνδράμει επίσης και τα μέλη ε, που ε, αντιμετωπίζουν αντίστοιχα δικήματα και να βοηθήσει και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα και να συνεργαστεί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και με τον είπα το εκπρόσωπο για τη σεξουαλική βία σε περίπτωση ενόπλων σειράξεων. Αύριο είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και θα ήθελα να ενθαρρύνω όλου του συναδέλφου να συνεργαστούν μαζί μου. Είμαι στη διάθεσή του ε, και στη διάθεσή σα για σχόλια, ακόμα και αν είναι επικριτική φύσεω, ε, για το σχέδιο γνωμοδότηση. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Μάισλες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Σιμάνσκι. Η έκθεση της ΑΦΕΤ, που είναι η βάση της νομοδότησης, είναι εκτενέστατη, αλλά στην παράγραφο 29 αναφέρεται σε γυναίκες και παιδιά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η γνωμοδότηση από την Επιτροπή μας γιατί πράγματι σε αυτή την Επιτροπή έχουμε ασχοληθεί με ακροάσεις, με θέματα τη σεξουαλική βία κατά των γυναικών, των παιδιών σε εμπόλεμες ζώνες και αυτό είναι κάτι το οποίο συχνά ε, συμβαίνει. Συμφωνώ με τη γνωμοδότηση εν πολλής. Θα κάνω μόνο τις εξής παρατηρήσεις που θα υποβάλω και ως τροπολογίες. Στο σημείο Β καταρχήν μου είναι σημαντικό να πούμε ότι η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται ως όπλο σε εμπόλεμες ζώνες κατά των γυναικών και των παιδιών Υπήρχε ε, μέσος σε πολλά σημεία, αλλά θα ήθελα να το αναδείξουμε και να το πούμε. Επίσης, στις παραγράφους 5 και 6 υπάρχει ε, μια έμεση μόνο και όχι άμεση αναφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οπότε απομονώνονται λίγο από το γενικότερο περιεχόμενο οι παραγράφοι αυτές γιατί πάντοτε αναφέρθηκε ε, η σχέση με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οπότε και εδώ θα πρέπει να υπάρχει η αναφορά, ιδιαίτερα ε, για να ενταχθεί στο κείμενο η παράγραφος 6. αλλά και η παράγραφος 5. Κατά τα άλλα, συμφωνώ. Ευχαριστώ. Σας κυρία Παπαδοπούλου τώρα. Ελπίζω να έχω το δικαίωμα να μιλήσω γιατί δεν είμαι τακτικό μέλος της Επιτροπής. Εκπροσωπώ τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα, του σοσιαλιστέ, ε, και ήθελα να θέσω ένα δικαστικό σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Σινκλέρ, διότι αν τα αναπληρωματικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα, μπορούν να είναι σκιώδη εισηγητέ. Ε, μάλλον το αγνοεί, αλλά έχει φύγει και δεν μπορεί να ακούσει την απάντησή μου. Έχω δικαίωμα να είμαι σκιώδη εισηγήτρια για αυτή την έκθεση. Συμφωνούμε λοιπόν με αυτή την έκθεση, τώρα την υποεξέταση έκθεση, ε, απολύτω, γιατί αναφερόμαστε στου βιασμούς, τους διωγμούς των γυναικών και των παιδιών ε, στις ένοπλες σειράξει και ναι στην Επιτροπή ΑΦΕΤ, στη βασική έκθεση που είναι και πάρα πολύ καλή αναφέρεται η ανάγκη να τονίσουμε ότι είναι χρήσιμη και η δική μας γνωμοδότηση και είναι χρήσιμος και σκόπιμο να εισαχθεί αυτή η ιδέα. Θα ήθελα στην έκθεση να μην αναφερόμαστε μόνο στα θέματα βίας που υφίστανται οι γυναίκες και τα παιδιά στις διεθνείς συγκρούσεις και ότι αυτό αναφέρεται στο σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ και προβλέπονται κυρώσεις. Προσωπικά θα ήθελα ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρουν τρόπους να εφαρμοστούν αυτά τα ψηφίσματα, να εφαρμοστούν αυτές οι Είμαι από την Κύπρο και έχω, είμαι πρόσφυγας και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη, ε, πώς είναι οι ζωές των θυμάτων. Ε, ξέρω τι γίνεται με τους πρόσφυγες, με τους αγνοούμενους. Έχουμε δει πολλαπλά ψηφίσματα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, αλλά δυστυχώς ε, υπάρχουν εδώ και χρόνια, αλλά δεν εφαρμόζονται. Πρόκειται για μια πολιτική φρασιολογία. Δεν, το θέμα μας δεν είναι να υγείρουμε μόνο τα ζητήματα. Ε, το θέμα είναι να ε, εφαρμοστούν ε, τα ψηφίσματα του ΙΕ και οι γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σχέση με το περιεχόμενο του σχεδίου θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι πολύ καλή έκθεση. Ίσως να υποβάλουμε και κάποιες τροπολογίες για να τονίσουμε την περαιτέρω τα είδη της σεξουαλικής βίας και να διευκρινίσουμε το ψυχολογικό τραύμα που Ευχαριστούμε κυρία Παπαδοπούλου. Τώρα ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μπέγκμαν, θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την Κομισιόν ΜΕΝ, αλλά δεν έχουμε σχόλιο. Ωραία. Τότε να ακούσουμε τον κύριο Σισμέσκη και πάλι τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλιά σας. Περιμένω και τις προτάσεις που μου αναφέρατε. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θέματα να αντιμετωπίσουμε, πολύ περισσότερα όπως αναφέρω εδώ, διότι είναι ευρύτατο το ζήτημα. Για μένα ως συντάκτη της γνωμοδότησης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ε, συμμετοχή από πολλές χώρες ε, ε, μειώνει, υποβαθμίζει το ρόλο του δικαστηρίου. Αυτά τα οποία συνέβησαν στη Ρωσία δεν θα πρέπει να μας αποτρέψουν, θα πρέπει να ασκήσουμε και άλλες πιέσεις. Η συμμετοχή της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας δεν θα δώσουν απαραίτητα την αποτελεσμάτικα που χρειαζόμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη δύναμή της και τις δυνατότητές της και για πολιτικούς και οικονομικούς στόχους φαίνεται να θυσιάζουμε τις αξίες μας και αυτό είναι σαφές παράδειγμα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τις ε, θετικές προκαταρκτικές σας απαντήσεις. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια και νομίζω ότι αυτό είναι απόδειξη ότι έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα κείμενο το οποίο θα είναι αποδεκτό από όλους. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιμένσκι. Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής. Δεν ακούμε δυστυχώς την πρόεδρο γιατί δεν μιλάει στο μικρόφωνο. 11 Οκτωβρίου νομίζουμε στην Επιτροπή ΑΦΕΤ θα ψηφιστεί η έκθεση ε, και στην Ολομέλεια θα ψηφιστεί τον Νοέμβριο του 2011 προφανώς. Eh, Περνούμε τώρα στο τελευταίο σημείο προσεχής συνεδρίαση. Σας είπα ήδη Στρασβούργο 15 Σεπτεμβρίου από τις 8.30 ε, μέχρι τις 10.30 και μετά στις ε, Βρυξέλλες ε, η συνεδρίασή μας στις 11 Οκτωβρίου και πρωί και απόγευμα. Ολοκληρώσαμε τώρα το, την μερίσια διάταξη. Καλό απόγευμα σε όλους.